start, nevertheless. It is far from the main building, therefore I think uh, some people are still on their way. Είμαστε μακριά από το κεντρικό κτίριο και νομίζω ότι κάποιοι ακόμη δεν έχουν φτάσει. Θα μιλήσω γερμανικά τώρα. Ordnung. Das ist nicht der Fall. Die... Τα πρακτικά των ε, δύο τελευταίων συνεδριάσεων ε, σα έχουν κατατεθεί. Σίγουρα δεν νομίζω να δεν θα υπάρξουν ε, αντιρρήσεις σε σχέση με την ημερήσια διάταξη. Για το γλωσσικό μας καθεστώς έχουμε κάποιες ελλείψεις. Εκτός από τα σουηδικά έχουμε όλες τις γλώσσες. Ω συνήθως. Η κυρία Μαγκόσα Κασλίντα είναι το νέο μέλος της ε, γραμματείας μας. Καλωσορίσατε, μπορείτε να σταθείτε λίγο όρθια για να σας δούνε. Έρχεστε από την Επιτροπή Γυναικών. Ε, καλή τύχη σας εύχομαι. Mit Ihnen streiten können, aber Βεβαίω, ε, μερικές φορές ε, έχουμε διαφωνίε, ε, αλλά όλα αυτά αφορούν την ουσία και κατά τα άλλα Σήμερα το πρωί έχω το εξή ε, πρόβλημα. Γύρω στι 10 ε, πρέπει να πάω σε μια άλλη συνεδρία. Θα επανέλθω βέβαια ο συνάδελφο κ. Ε, Φοντάνα. Αν βέβαια έχει έρθει εντωμεταξύ θα με αντικαταστήσει. Αυτήν την εβδομάδα ή τι τελευταίε εβδομάδε από την τελευταία συνεδρίαση είχαμε διάφορε τριμερείς διαλόγους το, ο τρίλογος η τριμερή συνάντηση Εράσμους για όλους την Περασμένη Δευτέρα είχαμε τον τελευταίο τριμερή διάλογο και στις 11 και 12 Μαρτίου είχαμε τον τελευταίο τριμερή διάλογο και προβλέπονται άλλοι δύο τριμερείς διάλογοι για το νέο πρόγραμμα για την ε, νεολαία. Κοιτάξτε, δεν θα συνεχίσω να διαβάζω γιατί μπερδεύτηκα. Είχαμε λοιπόν τρει τριμερεί διαλόγου. Πρώτα για την εκπαίδευση και για τεχνική φύσεω θέματα, για την ε, ε, νεολαία και για τον αθλητισμό και είχα την εντύπωση ότι το Συμβούλιο ε, ευχάριστα προσφέρει τη βοήθειά του και είχαμε τώρα μια πάρα πολύ καλή έκβαση της υπόθεσης. Οι συνάδελφοι μέχρι πρόσφατα ήταν πάντα παρόντες. καταρχήν συζητήσαμε για τους γενικούς στόχους, μετά ε, ασχοληθήκαμε με τη νεολαία και τον αθλητισμό σε πάρα πολλούς τομείς, επιτύχαμε μια μεγάλη προσέγγιση και επειδή το Συμβούλιο ε, επέδειξε πνεύμα συνεργασίας και η Κομισιόν. Όσον αφορά την εκπαίδευση και τον αθλητισμό, θέλω να σας πω ότι σχεδόν συμφωνήσαμε και απομένουν μόνο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ε, οριζόντιες επιτυχές του θέματος έτσι ώστε ε, να μπορούμε να ε, αντιδράσουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και τα παραθέσαμε αυτά μέχρι το τέλος. Ε, ας πούμε, ε, τις κατεξουσιοδότηση πράξεις ή τις εφαρμοστικές πράξεις, όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν είναι ιδιαίτερα επικοδομητικά. Εκείνο που δεν συζητήσαμε είναι το master loan, διότι το Συμβούλιο δεν έχει συμφωνήσει ακόμα επ' αυτού. Δεν μας έχει ενημερώσει κατά πόσον επιθυμεί κάτι τέτοιο ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε και προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε το Συμβούλιο και ίσως το θέμα αυτό να το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν μπορέσαμε να επιλύσουμε, είναι τα περίφημα brand names. Θα το εξετάσουμε αυτό σύντομα, αλλά πρέπει να σας πω ότι επί του θέματος αυτού ε, δεν υπάρχουν εμπόδια. Κατά τα άλλα, λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Την επόμενη Δευτέρα τη συνεδρίασή μα την αναβάλαμε διότι το Συμβούλιο δεν έχει λάβει ακόμα την εντολή. Την εντολή αυτή θα τη λάβει τέλη Μαρτίου έτσι ώστε να ε, συνεχιστούν διαπραγματεύσει στι 8 Απριλίου. Σε γενικέ λοιπόν γραμμέ, ο τριμερή διάλογο ε, προχωράει καλά. Στην επικοδομητική Ευρώπη μιλήσαμε επί του θέματο. Ε, στις 8 Φεβρουαρίου. Ε, τότε το Συμβούλιο δεν είχε ακόμα εντολή Κατόπιν τούτου, ε, ναι μεν ήμασταν παρόντες και συζητήσαμε, αλλά ε, η Ιρλανδική Προεδρία μόνο στις 6 Μαρτίου έλαβε την εντολή και αύριο το πρωί θα έχουμε τον πρώτο τριμερή διάλογο ε, που αφορά την δομή του προγράμματος, τον καθορισμό των στόχων, όπως επίσης και το ρόλο του παρατηρητηρίου και των Creative Desks όπως αποκαλούνται που το αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα κράτη-μέλη. Και κατόπιν έρχεται, αν θέλετε, το μεγάλο πρόβλημα, η Ευρώπη των πολιτών. Υπάρχει μια κατάσταση ε, η οποία λέει ότι θα πρέπει καταρχήν να υπάρχει συναπόφαση, αλλά δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Εμείς είπαμε ότι ε, θα συμπεριφερθούμε σαν να υπήρχε η συναπόφαση και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε όλες μας τις επιθυμίες στο Συμβούλιο. Κατά περίεργο τρόπο, ε, σε αντίθεση με όσα μου είχαν ήδη πει, το Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να προσεγγίσουν τη θέση μας, ίσως όχι από την αρχή. Αλλά ε, αφού ε, τους κάλεσα με τον κύριο Τάκουλα στο γραφείο μου χωρίς να χρειαστεί να τους ε, προσφέρω σαμπάνια κατορθώσαμε να επιτύχουμε αρκετά. Επιπρόσθετα σε αυτά που είχαν ήδη δεχτεί επιτύχαμε και τροποποίηση του κειμένου. Και τώρα λοιπόν θα προσπαθήσουν το όλο θέμα να το διευκρινίσουν με την Κορεπέρ. Και αν η Κορεπέρ συμφωνήσει πρέπει να συναντηθούμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Κατά πόσον θα επιμείνουμε στα νόμιμα δικαιώματά μας ή μήπως ε, χάρη των ε, χριστών είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε τις δικές τους απόψεις. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και πάλι. Όλα λοιπόν βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους οι οποίοι είναι πάντα παρόντες και οι οποίοι στις προκατακτικές συζητήσεις είναι ανοιχτοί για αλλαγές, αλλαγές και τροπολογίε που ενδεχομένω έχουν καταθέσει και οι ίδιοι και είναι πρόθυμοι να τι εντάξουν σε συμβιβαστική πρόταση με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Αυτή λοιπόν είναι η έκθεση που θέλατε να ακούσετε σχετικά με, τις, με τους τρεις τριγωνικούς διαλόγους. Το πρόγραμμα Creative Europe ε, θα είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει με το πρόγραμμα αυτό και δεν είμαι ακόμα σίγουρη κατά πόσον λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε πόσα χρήματα θα πάρουμε, κατά πόσον στο πλαίσιο του προγράμματος Creative Europe μπορούμε να συζητήσουμε και το θέμα των ε, δανείων. Ε, τα δάνεια αυτά θα δίδονται υποτίθεται από χρηματοψηφιακά ιδρύματα σε διάφορα κράτη-μέλη. Αυτά είχα να σας πω. Δεν ξέρω αν έχετε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Από ό,τι βλέπω δεν έχετε και πάμε στο σημείο υπαριθμών 4 της ημερήσιας διάταξης. Ε, έχουμε αναθέσει μια έκθεση στον συνάδελφο Αλφόνση που αφορά στις ε, υποαπειλή ε, τις γλώσσες που αντιμετωπίζουν την ε, απειλή της εξαφάνισης. Ε, κοιτάξτε, εδώ δεν πρόκειται για γλώσσες ε, γιατί το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή μας κατά το παρελθόν και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στις ε, τροπολογίες. Οι γλώσσες μειονοτήτων είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση. Αυτό παρακαλώ να το έχετε κατά νου στο βαθμό που θα καταθέσετε τροπολογίες. Γιατί δεν θα επιτρέψω καμία τροπολογία που θα ακολουθεί λάθος κατεύθυνση. Γιατί αυτό θα μας οδηγήσει σε περιττή συζήτηση για ένα θέμα που Ήδη το έχουμε εξετάσει και κλείσει αν θέλετε. Από ό,τι πληροφορήθηκα έχουμε 3.000 γλώσσες ε, οι οποίες πραγματικά απειλούνται με εξαφάνιση και γι' αυτό λοιπόν τον λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ε, αυτό ε, το θέμα αφορά τις τις πολιτιστικές μας ταυτότητες και νομίζω ότι εδώ πρόκειται για μια πολύ καλή ιδέα. Είχαμε μια ε, ομάδα ε, που συστήθηκε αποτελούμενη από πολλές ε, πολιτικές ομάδες. Ο Σαλφόνση προσφέρθηκε και σήμερα έχουμε και ε, πολλούς προσκεκλημένους. Τον κύριο Μόσλι, ο οποίος ε, είναι ο ε, αρχισυντάκτης του Παγκόσμιου Χάρτη των Υποεξαφάνιση Απειλούμενων Γλωσσών. Είναι ένα πρόγραμμα, αρμόδιο, αρμόδιο για το πρόγραμμα είναι η UNESCO και θα λάβει πρώτος τον λόγο. Έχουμε την Ιτσιφό, εκπρόσωπο της Γραμματείας ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, για τις ε, γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ κυρία μου ότι πρόκειται εδώ για γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση. Σας παρακαλώ να μην μου δημιουργήσετε το πρόβλημα που μόλις πριν από λίγο έκλεισα. Κατόπιν τον κύριο Φερνάντο, ο οποίος ασχολείται με την προβολή της γλωσσικής πολυμορφίας και έχουμε και τον Price Jones, επικεφαλής του APLD που είναι το δίκτυο για την προαγωγή της γλωσσικής πολυμορφίας και θα καταθέσει ένα σημείο, μια εισήγηση για αυτό το θέμα των γλωσσών που απειλούνται με εξαφάνιση. Μέχρι τις 11 έχουμε χρόνο για το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στον κύριο Αλφόνση για να μας παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του και Κατόπιν όλοι οι εμπειρογνώμονες έχουν στην αρχή 10 λεπτά, ε, θα ακολουθήσουν ερωταπαντήσεις και θα ε, δοθούν οι απαντήσεις των εμπειρογνωμόνων στα θέματα που θα έχουν τεθεί. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, κύριε Αλφόνση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα αφήσω μάλλον ε, να μιλήσουν οι προσκεκλημένοι μας, ε, αλλά εν συντομία να σας πω ότι ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες που ανέκαναν στη μέρη σε διάταξη αυτό το θέμα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη. μου. Πρόκειται για την πολιτιστική μας κληρονομιά, τη διατήρηση, τη διασφάλιση της ε, σε μια περίοδο όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι ανησυχητική κατάσταση και οι γλωσσικές κοινότητες ε, που έχουν σκληροδότημα μια ευρωπαϊκή γλώσσα τελούν σε απόγνωση ενίοτε και ε, πρέπει να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο πρέπει να αποφύγουμε ανεπανόρθωτες ζημιές και απώλειες του πολιτιστικού κληροδοτήματος αυτού. Ε, πρώτα απ' όλα όταν εργαζόμαστε για αυτές τις ε, ε, κοινότητες ε, υπερασπίζουμε και την ψυχή της Ευρώπης και βοηθούμε την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από τη γλώσσα υπάρχουν και οι πολιτιστικές πρακτικές που συνδέονται ούτως ή άλλως με κάθε γλώσσα από τις εικαστικές τέχνες, γαστρονομικές περιπέτειες. Πρόκειται για πολιτιστικά κοιτάσματα που τροφοδοτούν την κληρονομιά μας στην Ευρώπη. Αφήνω λοιπόν το λόγο στους κλειμένους μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Αλφόνση. Ε, ο κύριος Μόσλι θα πάρει το λόγο. Παρακαλούμε. Thank you. Um, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη τιμή για μένα αλλά και μεγάλη χαρά. Ε, βρίσκομαι εδώ να σας μιλήσω για τον Άτλαντα, τον γλωσσών που κινδυνεύουν, ε, έναν άτλαντα τη UNESCO. Βλέπετε ε, την έκδοση και έχουμε και έναν οδικό χάρτη. Ελάτε μετά να σας δείξω τον άτλαντα αυτό. Προς το παρόν όμως θα ήθελα να σας εξηγήσω πώς ε, καταρτίστηκε και από πού ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Πώς ορίζει η UNESCO τις γλώσσες που απειλούνται. Σε τι κατάσταση πρέπει να είναι μια γλώσσα για να πάρει μια θέση σε αυτό το χάρτη, σε αυτό τον Άτλαντα. Ένα ορισμό θα ήταν ότι μια γλώσσα κινδυνεύει με εξαφάνιση όταν δεν τη μαθαίνουν πια τα παιδιά. Αλλά για να ορίσουμε έτσι πιο συγκεκριμένα την έννοια αυτή, θα πρέπει να εξετάσουμε κάποιου παράγοντε. Πρώτα απ' όλα, τον απόλυτο αριθμό μιλούντων τη γλώσσα, τη διαγενειακή μετάδοση της γλώσσας, την αναλογία των ομιλητών μέσα στο πληθυσμό τη στάση των μελών της κοινωνίας απέναντι στη γλώσσα τους, τη διαθεσιμότητα υλικών για την εκπαίδευση, για τον αλφαβητισμό, τον εγγραμματισμό, τους τομείς στους οποίους χρησιμοποιεί τη γλώσσα, την ανταπόκριση σε νέους τομείς, σε νέα μέσα, μίντια, το είδος, την ποιότητα των εγγράφων, της τεκμηρίωσης και βέβαια την κρατική και τη θεσμική στάση και πολιτικές. Μεταξύ αυτών την επίσημη κατάσταση, το επίσημο καθεστώς και την επίσημη χρήση αυτής της γλώσσας. Όλοι από κοινού αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν ε, στο κατά πόσο είναι πιθανό να κινδυνεύει μια χώρα ε, με εξαφάνιση ή όχι. Το 1996 υπό τον Στίβεν Βούρμ, τον καθηγητή Στίβεν Βούρμ στο Αυστραλιανικό Πανεπιστήμιο ε, καταρτίστηκε για πρώτη φορά. Ο Άτλαντας και περιλάμβανε 600 ε, γλώσσες. Είχαμε 53 σελίδες και 12 χάρτες. Δεύτερη έκδοση, 2001, με τον ίδιο καθηγητή ε, συντάκτη, ολοκληρώθηκε μάλιστα λίγο πριν αποβιώσει καθηγητή σε Βούρμα. Σε αυτή την έκδοση ε, που είχαν συμμετάσχει και μια εθνική ομάδα εμπειρογνώμων, περιγράφεται η κατάσταση, συνοδεύεται δηλαδή ε, ο κάθε χάρτη από συγκεκριμένη περιγραφή. Έχουμε τι γλώσσε που απειλούνται υπό εξαφάνιση με ένα σύστημα ε, έγχρωμων κωδικών, χρωματικών κωδικών. Το ίδιο έχουμε και εμεί ακολουθήσει. Από 600 είχαν πάει στις 800 ε, είχαμε 90 σελίδες ε, κείμενο, 14 χάρτες. Πάλι όμως δεν ήταν πλήρης ο Άτλαντας. Χάρη στην χρηματοδότηση της νορβηγικής κυβέρνησης, ε, αρκετά γενναιόδορη, καταφέραμε να επεκτείνουμε αυτό το project υπό διάφορους τρόπους για, το νέο, για την νέα έκδοση. Σε δύο μορφές πια, μία ψηφιακή, online, εκδόση που μπορεί κανείς να τη δει με την, από την ιστοσελίδα της UNESCO και την έντυπη μορφή, αυτή που έχω φέρει μαζί μου. Η ψηφιακή εκδοχή ε, λανσαρίστηκε το Φεβρουάριο του 2009 στο Παρίσι την ε, Διεθνή ημέρα μητρικών γλωσσών και η έντυπη μορφή ένα χρόνο μετά δημοσιεύτηκε και στα ισπανικά και στα γαλλικά. Τρει δηλαδή σε τρει γλώσσε ε, κυκλοφορεί ο Άτλαντα αυτό. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα ότι τώρα είναι προσβάσιμο για όλου του χρήστε μέσω του διαδικτύου. Άρα, αν υπάρχουν παραλήψει, παροράματα, ε, διορθώσει που χρειάζεται να γίνουν, όλα αυτά μπορούν εύκολα ε, να συμβούν στην ηλεκτρονική εκδοχή και να μπουν και οι διάφορε τροποποιήσει σιγά-σιγά μετά και στην έντυπη στον έντυπο Άτλαντα. Περιλαμβάνονται τώρα 2.500 γλώσσες, ή μάλλον παραπάνω. Ίσως δηλαδή πάνω από το 1 τρίτο ε, των γλωσσών παγκοσμίω. Μία γλώσσα κάθε λίγες εβδομάδες σβήνει, έτσι μας λένε οι ειδικοί, πεθαίνει. Η συντακτική ομάδα πρέπει να αποφασίσει να συμπεριλάβει και κάποιες γλώσσες που ε, εξαφανίστηκαν πρόσφατα. 230 περίπου από τις χώρες που περιλαμβάνονται εξαφανίστηκαν από το, ε, από το 1950 και μετά. Δύο γενιές ε, ε, έχουν χάσει γλώσσες θα λέγαμε. Από τότε που ιδρύθηκε η UNESCO δηλαδή. Πριν οι έντυποι χάρτες είχαν ένα χρώμα μόνο και είχαν ε, τυπωθεί στη σχετική κλίμακα, δεν είχαν όμως απογραφικά στοιχεία και πολύ λίγοι δείκτες υπήρχαν, δηλαδή κάποια σημαντικά γεωγραφικά ε, στοιχεία και κάποιες πόλεις. Τώρα, βέβαια, δεν έχουμε υπερφορτωμένους με γεωγραφικά στοιχεία Άτλαντες, βασιζόμαστε όμως στο Google Maps. Δεν θέλουμε να μπερδεύεται ο χρήστη. θέλουμε να μπορεί να δει εύκολα ε, πού ομιλείται η κάθε γλώσσα, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη γεωγραφική λεπτομέρεια και μπορεί κανείς να ζουμάρει ε, με διαφορετικές κλίμακες στην ηλεκτρονική έκδοση, άρα μπορεί πολύ εύκολα ο χρήστη να τοποθετηθεί και στην online έκδοση μπορεί κανείς να επιλέξει τη γλώσσα κλικάροντας το σύμβολο. Μια γλώσσας και να δει τι στοιχεία υπάρχουν διαθέσιμα για την κάθε μεμονωμένη γλώσσα. Μπορείτε και εσείς να ε, δοκιμάσετε. Δεν έχω οθόνη ε, μπροστά μου, πολύ απλό. είναι το site www.unesco.com.org και μετά θα μπείτε στην και μπορείτε να δείτε τον Άτλαντα τι δεδομένα θα είχατε. Το όνομα, ε, αν υπάρχει κάποια αναλεκτική ονομασία, ε, κώδικα του ISO 63 κάθετος 3, 369 κάθετος 3, αλλά ε, αν αναγνωρίζεται ε, ξεχωριστά, μια ως ξεχωριστή γλώσσα, πώς ποσοτικοποιείται αυτό ε, μια γλώσσα. Είναι, υπάρχουν κάποια σημαντικά κριτήρια, γιατί αφενός μια γλώσσα μπορεί να έχει πολλά ονόματα, πολλές ονομασίες. Μπορεί να μιλάει επίσης κάποιος για διαλέκτους αυτής της γλώσσας και απ' την άλλη μπορεί πολλές γλώσσες να έχουν το ίδιο όνομα. Άρα έχουμε τον κώδικα, τον κωδικό που θα τις ξεχωρίσει και θα τους δώσει της καθεμιάς μια ταυτότητα. Έχουμε περιοχές υπηρετικές και για κάθε περιοχή οι δικοί μας έχουν εργαστεί πάνω στις περιοχές και δίνουν τα στοιχεία. Έχουμε έναν web editor ε, στα γραφεία, στα κεντρικά της UNESCO στο Παρίσι, ο οποίος ε, μπορεί να δώσει και τις νοδευτικές πληροφορίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις γλώσσες, οι οποίες έχουν ευρετηριαστεί και καταγραφηθεί με αλφαβητική σειρά. Μπορεί κανείς να τις δει ε, κάνοντας scroll down ε, σε ένα μενό. Και βλέπουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, μπορεί να εμφανίζεται να εμφανίζονται πολλές γλώσσες ή η ίδια γλώσσα σε περισσότερες της μιας χώρες. Μπορεί κανείς να, να δει και τον κατάλογο, το index και στην έντυπη μορφή έχει κανείς τον κωδικό ISO. Κάποιες φορές όμως οι ειδικοί ε, διαφωνούσαν με τους κωδικούς, είτε γιατί θεωρούσαν ότι εφαρμόζονται πολύ ευρέως, σε πολλές γλώσσες δηλαδή, ή πολύ στενά. Οπότε δεν εντοπίζονται σωστά, δεν ταυτοποιούνται σωστά κάποιες διάλεκτοι, κάποιες γλώσσες. Οπότε ε, γίνονται κάποιες διορθώσεις στον επίσημο κατάλογο κωδικών και κάποιες φορές βλέπουμε ότι χρειάζονται νέοι κωδικοί ή κάποιοι παλιοί κωδικοί θα πρέπει να επαναποδοθούν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για τη χαρτογράφηση γλωσσών στον αυτό είναι ότι γλώσσες δείχνονται με ε, σημεία, όχι με πολύγωνα. Άρα έχουμε ένα στάνταρτ μέγεθος για την κάθε γλώσσα. Ε, γιατί ε, είναι απλό. Αν είχαμε πολύ μικρά κουκίδες θα μπορούσαν να χαθούν, ενώ αν είχαμε μεγαλύτερες κουκίδες μπορεί να σβήνονταν από αυτές τις κουκίδες κάποιες μικρότερες, να τις κάλυπτε δηλαδή μεγαλύτερη κουκίδα ούτε πολύ να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ούτε άλλα σχήματα τα οποία να ε, εκπροσωπούν την περιοχή στην οποία μιλείται μια γλώσσα. Γιατί τελικά δεν θα είχε κάποιο νόημα και θα δημιουργούσε προβλήματα, απορίες. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίσαμε την πρόκληση να βάλουμε αυτή την κουκίδα, τη στάνταρτ κουκίδα ε, για τις ε, γλώσσες. Αν είναι διασκορπισμένοι χρήστε τώρα μια γλώσσα σε μια ευρύτερη περιοχή, σε Βηρία ή σε μέρη τη Βορειοαμερική για παράδειγμα, έχουμε και άλλο πρόβλημα και αν υπάρχουν μεταξύ αυτών και άλλες γλώσσες, άλλε άλλες δηλαδή, άλλα σημεία, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο πολλές κουκίδες. Προσπαθήσαμε να είμαστε οικονόμοι ε, και πρέπει έτσι με, με λογική και ε, οικονομία ε, να αποδίδουμε όλα αυτά τα σημεία, αυτές τις κουκίδες πάνω στους χάρτες. Κάναμε λοιπόν αυτή την απονομή, δώσαμε ένα, ένα χρώμα, πηγαίνοντας από το, από το κίτρινο μέχρι το μαύρο, ανάλογα με τη σοβαρότητα, με του κινδύνου που αντιμετωπίζει μια γλώσσα να εξαφανιστεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δεγενειακή ε, μετάδοση, εάν είναι αδιάλειπτη, τότε δεν βλέπουμε τις χώρες αυτές στο ε, στον Αν απειλείται η διαγενειακή μετάδοση, ε, μόνο τότε αρχίζει να φαίνεται. η πολυγλωσία μπορεί να αναφέρεται. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε ε, πολυγλωσία ή κάποιες γλώσσες επικρατούν. Όλα αυτά τα παρακολουθεί η Συντακτική Επιτροπή και οποιαδήποτε αλλαγή υπάρχει την εντοπίζει. Ε, έχουμε μια άλλη κατηγορία. Έχουμε λοιπόν πρώτα safe, μετά vulnerable, ευάλωτη. Μπορεί δηλαδή να ομιλεί τη γλώσσα από τα παιδιά αλλά στο σπίτι όχι επισήμω, αλλά στο σπίτι. Μετά έχουμε έναν επόμενο βαθμό, definitely endangered. Αν δηλαδή η γλώσσα δεν μαθαίνεται πια ε, ως μετρική γλώσσα, ούτε διδάσκεται και στο σπίτι. Και οι νεαρότεροι ε, ομιλητέ τη είναι οι γονεί. Εκεί ε, έχουμε το πρόβλημα. Μετά, severely endangered, όταν μόνο οι γονεί και οι παλιότερε γενιέ ε, μιλούν τη γλώσσα, ή μάλλον οι γονεί μπορεί να την καταλάβουν, αλλά όχι να την μεταδώσουν στα παιδιά του. Επόμενη κατηγορία, critical endangered που είναι το, το δεύτερο πιο σκούρο χρώμα, δηλαδή αυτοί που μιλούν ε, την ε, γλώσσα ε, είναι οι παππούδες ή προπάποι και εκεί πλέον δεν μιλείται σχεδόν καν η γλώσσα και δεν έχει κάποιος έναν συνομιλητή εύκολα για να τη μιλεί. Και όπως είπα μετά τελευταία κατηγορία extinct, ήδη εξαφανιστεί σας γλώσσες δηλαδή, μαύρο χρώμα, αν κανείς δεν τη μιλά αυτή τη γλώσσα. Σα είπα ότι οι συντάκτες αποφάσισαν να συμπεριλάβουν ε, γλώσσες που έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία 60 χρόνια. Αυτό για μας είναι το πιο επίμαχο ζήτημα και δημιούργησε τις πιο πολλές συζητήσει μετά την ε, δημοσίευση του Άτλαντα. Πολλά ακόμα θα μπορούσα να πω. Ε, the, of the... Θα σας πω όμω σε ποια φάση τώρα τη δουλειά μας βρισκόμαστε. Είναι ενδιαφέρουσα το Ίδρυμα για τις ε, υποεξαφάνιση γλώσσες, ένα ίδρυμα Μέδρα τη Βρετανία, το ανάθεσε λοιπόν η UNESCO αυτού του Ιδρύματος να ε, προβεί σε ένα feedback από τους χρήστες. Ένα feedback το οποίο εδώ και δύο χρόνια, ή μάλλον όχι, τέσσερα χρόνια από όταν ε, δημοσιεύτηκε online ο Άτλαντας. Λαμβάνεται λοιπόν εδώ και τέσσερα χρόνια αυτό το feedback. Αρχικά ε, είχαμε αρκετά σχόλια τη μέρα, υπήρχε μεγάλο ε, ενθουσιασμό. Τώρα έχουμε κανένα δύο σχόλια τη βδομάδα. Και βέβαια πρέπει να ελεγχθεί η ακρίβεια των ισχυρισμών, αντιχειρισμών κτλ. Αυτό είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ ε, χρονοβόρα, δύσκολη, γιατί πρέπει να γίνει με ακρίβεια και με σοβαρότητα. Πρέπει να εντοπίσουμε ε, τους δείκτες, να τους κατατάξουμε στην κλίμακα, να δούμε ποιοι ε, είναι οι ομιλητές, πόσοι αν είναι μια γλώσσα, αν είναι μια διάλεκτος, βιβλιογραφικές πηγές να ζητηθούν, εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγματο χάρη και ανέκδοτα για το ε, αν μιλούν εθνοπολιτικές δηλώσεις από εκπροσώπους ε, μειονοτήτων που θέλουν να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους, από αυτούς παίρνουν πολύ feedback και γενικά ζητήματα που αφορούν κριτήρια που σχετίζονται με την UNESCO. Θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα. Αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσω τώρα. Και θα μπορέσω να σας διαφωτίσω περαιτέρω απαντώντας τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, θα ήταν ε, βέβαια πολύ πιο εύκολο να σας παρακολουθήσει κανείς. Αν είχατε και κάποιες διαφάνειες να μας προσβάλλετε, κάτι, κάποια, ένα PowerPoint. Κοιτάξτε, έχω PowerPoint. Ε, α, στην αρχή έπρεπε να μας το πείτε αυτό αποφάσισα να μην το δείξω, να μιλήσω απλά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας ε, είπατε. Έχουμε ε, τώρα ε, την εκπρόσωπο από το Συμβούλιο της Ευρώπης που είναι αρμόδια για την προστασία των τον κύριο, με συγχωρείτε, τον κύριο που είναι αρμόδιος. Πότε ρωτάμε, μετά ή τώρα, μετά. Good morning. Καλημέρα σας. Εγώ θα εστιάσω την παρουσίασή μου στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για Περιφερειακές Γλώσσες Μειονοτήτων. Αυτός ο χάρτης είναι ο, η μόνη συμφωνία που υπάρχει στον κόσμο που αφορά στην προστασία ε, γλωσσών ε, παραδοσιακών μειονοτήτων. Πρέπει να πούμε ευθύ εξ αρχής ότι ο χάρτης δεν χρησιμοποιεί τον όρο γλώσσες ε, απειλούμενες με εξαφάνιση. Παρόλα αυτά όμως γίνεται αναφορά σε ιστορικές γλώσσες μειονοτήτων της Ευρώπης. Ορισμένες εξ αυτών πράγματι αντιμετωπίζουν την επιλή της εξαφάνισης. Όσοι συνέταξαν αυτό το χάρτη είχαν ε, μια ε, καινοτόμο προσέγγιση και από την άλλη προσφέρεται στο χάρτη μια πραγματική ευελιξία. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν ε, σε όλες τις γλώσσες ανάλογα με την κατάσταση. Οι περιφερειακές γλώσσες ή οι γλώσσες μειονοτήτων ορίζονται ως γλώσσες που χρησιμοποιούνται μέσα σε μια συγκεκριμένα περιφέρεια ενός κράτους και βέβαια αυτό αυτή η μειονότητα αριθμητικά είναι πολύ λιγότερη από τους υπόλοιπους πολίτες. Δεν περιλαμβάνονται βέβαια διάλεκτοι της επίσημης γλώσσας ή διάλεκτοι των μεταναστών. Ο χάρτης σήμερα αποτελείται από 25 μέρη, 16 ε, είναι από κράτη-μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν άλλα 11 όμως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν επικυρώσει το χάρτη. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και άλλα κράτη που και αυτά δεν έχουν επικυρώσει, όμως ε, για ορισμένες εξ αυτών των χωρών υπάρχει μια δέσμευτο Συμβούλιο της Ευρώπης για επικύρωση. Και στην περίπτωση των κρατών που πρόκειται να γίνουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής σε πράγματι τους έχει ανακοινωθεί και η υποχρέωσή τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαναγνωρίσει τη σημασία του χάρτη ε, όσον ε, αφορά τις υποχρεώσεις σε ένα ψήφισμα του 2003 και το ψήφισμα αυτό ορίζει τον χάρτη ως το ε, νομικό σημείο αναφοράς για αυτές τις γλώσσες. Όπως σας είπα ήδη ευθύς εξ αρχής, ο χάρτης είναι ένα καινοτόμο νομικό εργαλείο. Σε αντίθεση με άλλες συμβάσεις, ο χάρτης αυτός δεν εστιάζει στα δικαιώματα των πολιτών, αλλά στην προαγωγή των περιφερειακών γλώσσων, γλωσσών μειονοτήτων. Και έτσι λοιπόν τα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προάγουν αυτές τις ε, περιφερειακές γλώσσες των μειονοτήτων. Η προσέγγιση του χάρτη είναι αυτές οι περιφερειακές γλώσσες ε, να αποκτούν μια κοινωνική λειτουργία, κάτι που υπήρχε για πολλές εξ αυτών στο παρελθόν, έτσι ώστε ε, να παραμένουν ζωντανές οι γλώσσες. Εξάλλου υπάρχει υποχρέωση ε, να προάγονται αυτές οι γλώσσες στη δημόσια ζωή, δηλαδή στην εκπαίδευση, στα δικαστήρια, στη διοίκηση, στον πολιτισμό, στην οικονομική και κοινωνική ζωή, όπως επίσης και στην διασυνοριακή συνεργασία. Ο χάρτης είχε ως στόχο να καλύψει διάφορες γλώσσες στην Ευρώπη και ο τρόπος ε, με τον οποίο το κάνει αυτό το χάρτη συμβάλλει στο μοναδικό του χαρακτήρα. Ε, διαιρείται σε δύο μέρη όσον αφορά τις υποχρεώσεις του και υπάρχουν αρκετές αρχές στο δεύτερο τμήμα που αφορούν σε όλες τις περιφερειακές γλώσσες μειονοτήτων σε ένα κράτος. Κατόπιν, στο τρίτο τμήμα υπάρχει μία σειρά συγκεκριμένων υποχρεώσεων ότι τα που επιλέγουν τα κράτη ε, τις γλώσσες όπου ισχύουν αυτά τα μέτρα και υποχρεώσεις και επίσης επιλέγουν για κάθε γλώσσα τα μέτρα ε, τα οποία θα εφαρμόσουν. Τα μέτρα λοιπόν αυτά που αναφέρονται στο τρίτο τμήμα του χάρτη ακολουθούν τα εξή ε, παραδείγματα. Τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών των μηνοτήτων, απλά δηλαδή διδασκαλία. Δεν προβλέπεται να υπάρχει ε, τηλεοπτικό πρόγραμμα σε αυτή τη γλώσσα της ε, μειονότητας. Η, όσον αφορά τη χρήση της ε, γλώσσας σε επίπεδο διοίκησης παράλληλα με την επίσημη γλώσσα, πράγματι γίνονται αποδεκτές ε, αποδεκτά κάποια αιτήματα από πλευράς ε, μελών αυτής που χρησιμοποιούν αυτή την ε, γλώσσα των νοτήτων. Ο χάρτης προβλέπει μια ευελιξία. Ο χάρτης προστατεύεται με ένα μηχανισμό ελέγχου. Υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων που ελέγχει πως ο χάρτης αυτός εφαρμόζει σε διάφορα κράτη-μέλη και ο μηχανισμός καταθέτει και συστάσεις. Με βάση λοιπόν τη δουλειά των εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης καταθέτει συστάσεις στα κράτη-μέλη. Σήμερα ο χάρτης καλύπτει 84 γλώσσες που χρησιμοποιούνται από 206 ομάδες, μειονότητες. Ανάμεσα στις γλώσσες αυτές υπάρχουν ε, με πάρα πολλούς γλώσσες, με πολλούς ομιλητές. Ας πούμε, τα καταλανικά ή μία γλώσσα μειονότητα ε, στην Κύπρο που έχει σχέση με τα αραβικά προστατεύονται από την χάρτη. Στην Σλοβακία τα ουγγρικά προστατεύονται από τον χάρτη και έχουμε τα κροατικά, τα βουλγαρικά και τα πολωνικά που επίσης καλύπτονται από τον ε, χάρτη όμως μόνο όσον αφορά τη διδασκαλία της ε, γλώσσας. η δική μας Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχει συστήσει πρόσφατα να ληφθούν μέτρα για να ε, ε, διδαχθούν κυρίως τα εβραϊκά σε όσους τα επιθυμούν. Η Φινλανδία και αυτή έχει λιγότερο επίσημες γλώσσες, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει και η μειονότητα Σάμι, ε, η οποία και αυτή διδάσκεται στα, στην χώρα αυτή. Η τελευταία όμως εκδοχή αυτής της γλώσσας των νομοδιότητων έχει μόνο 200 ομιλητές. Έχουμε πολλές γλώσσες με περιορισμένο αριθμό ομιλητών. Στη Γερμανία, ας πούμε, ε, η Γερμανία μόλις τα τελευταία δέκα χρόνια έχει προσυπογράψει το χάρτη και γι' αυτό λοιπόν βλέπει κανείς ε, πώς έχει εξελιχθεί μια γλώσσα, ε, γλώσσες μειονοτήτων. Έχω ξεκινήσει από την απλή διδασκαλία και φτάνουν στην σημερινή μορφή όπου πραγματικά διδάσκονται και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπό την επιρροή λοιπόν του χάρτη βλέπουμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη, ίσως να μην είναι ιδανική, αλλά υπάρχει μια εξέλιξη. Υπάρχουν πολλές μορφές Βελτίωση βελτιώσεις όσον αφορά τη γλώσσα και οι βελτιώσεις αυτές αποδίδονται στο χάρτη. Ε, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε γλώσσες ε, ε, που δεν προστατευόντουσαν στο παρελθόν. Παραδείγματο χάρη τα σλοβενικά στη Γερμανία ή τα αραβικά στην Κύπρο. Έχει επίσης έχουν επίσης ε, υπάρξει και κάποιες γλώσσες μειονοτήτων που προστατεύονται ας πούμε στην ε, Ολλανδία, στο Σλέσβικ holstein στη Γερμανία. Εκεί υπάρχει και μια ε, γλώσσα της Βόρεια Φρίσλαντ, όπω λέγεται, που προστατεύεται από το χάρτη και άλλε όμω γλώσσε μειονοτήτων προστατεύονται στη Νορβηγία και αλλού. Υπάρχει μια μεγάλη πληθώρα γλωσσών που προστατεύονται από το χάρτη. Ο χάρτης αποτελεί ένα επαρκές εργαλείο για την προστασία όλων των γλωσσών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Λέει η Πρόεδρος, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα δίλημα όσον αφορά και πάλι τον διαχωρισμό, τον υποξαφάνιση απειλούμενων γλωσσών και των γλωσσών των μειονοτήτων. Χαίρομαι που υπάρχει αυτός ο χάρτης ε, που προστατεύει μια γλώσσα σε πολλές χώρες που ήταν γλώσσα των γηγενών και πλέον σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι οι γηγενείς έχουν τη δυνατότητα και να μάθουν και να μιλήσουν αυτή τη γλώσσα. Ας πούμε στα Βαλκάνια και εκεί προσπαθούμε τον χάρτη των Ηνωμένων Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το γλωσσικό να τον κάνουμε αποδεκτό. Θα αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Στη Σερβία, παραδείγματο χάρη, στην, ε, στη Βοηβοδίνα, η οποία στο κοινοβούλιο είχαν πάντα έξι γλώσσες. Στη Μακεδονία, άλλο παράδειγμα, τα αλβανικά ποτέ δεν μεταφράζονται. Τώρα όμως είναι επίσημη γλώσσα τα αλβανικά στο κοινοβούλιο της Μακεδονίας. Βλέπουμε λοιπόν πως ε, υπάρχουν προσπάθειες ε, που σχετίζονται άμεσα με την ε, πολιτιστική μας ταυτότητα. Όμως αυτές δεν είναι γλώσσες που απειλούνται από εξαφάνιση, είναι περισσότερο γλώσσες των μειονοτήτων. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, σχετικά με, το, με τη συμπερίληψη αυτών των γλωσσών στις δικές μας τις ε, συστάσεις. Επόμενος ε, ομιλητής από το Δίκτυο για την Προβολή της Γλωσσικής Πολυμορφίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω που προσκαλέστε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προώθηση της Γλωσσικής Πολυμορφίας για να σας παρουσιάσουμε το έργο μας. Το NPLD εδώ και 7 χρόνια λειτουργεί. Το 2006 ε, είδαμε ότι υπήρχε ένα κενό σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπωση των λεγόμενων συνταγματικών περιφερειακών ε, γλωσσών ή γλωσσών μικρών κρατών. Και έτσι γεννήθηκε το δίκτυο NPLD. Η δομή του είναι, έχει μία προεδρία η κυρία Ντεφρίες, υπουργό Οικονομικών και Πολιτικών της, ε, και της Επιτροπής της ε, περιοχής του Φρίσλαντ είναι η πρόεδρος. Έχουμε από ε, την Καταλωνία, από το Φόλτινγκ της Φιλανδίας, έχουμε και διευθυντή εκτελεστικό, έχουμε τους συμβούλους μας, τους διαχειριστές των προγραμμάτων, έχουμε στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παίρνουμε κάποια ε, ενίσχυση από το πρόγραμμα διαβίου μάθηση. 138.000 ευρώ ετησίω παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα διερωτηθείτε γιατί οι συνταγματικέ περιφερειακέ γλώσσε ή γλώσσε μικρών κρατών ε, είναι το αντικείμενο και γιατί όχι περιφερειακές γλώσσες ή απειλούμε εξαφάνιση ή μηνωτικές γλώσσες. Κάτι εντελώς διαφορετικό, όπως είδαμε και πριν παρουσιάσεις. Θα σας πω πολύ απλή απάντηση. Εμείς στο NPLD ασχολούμαστε με διαφορετικές γλώσσες, που είναι από γλώσσες ε, επίσημες, επίσημες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι ε, τα Ιρλανδικά ή τα αστωνικά, σε γλώσσες που είναι επίσημα αναγνωρισμένες σε κάποιες περιφέρειες των κρατών μελών, όπως είναι τα Γαλλικιακά, τα Βασκικά, ισπανικά, τα καταλανικά μεταξύ άλλων, ή γλώσσες που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, που αγωνίζονται να αναγνωριστούν επισήμω. όπως το οξιτάνικα, τα βρετανικά ή και τα κορσικά ενδεχομένω. Κρατικές λοιπόν γλώσσες, περιφερειακές, γλώσσες που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, μενοτικές, διάφορες ομάδες, ε, ε, ετερόκλητες ε, όλες αυτές οι κατηγορίες το Ιρλανδικά που είναι ε, επίσημη γλώσσα, ομιλούνται από 77.000 ανθρώπους ε, μόνο, ενώ 10 εκατομμύρια περίπου μιλούν καταλανικά. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τι μπορούν να έχουν κοινό όλες αυτές οι γλώσσες από τα σκανδιναβικές χώρες, το Σουηδικό δηλαδή για παράδειγμα, ή τα Κορσικά, στην, ε, μιλάμε πλέον για την Νότια Ευρώπη, ή στην Ανατολική που έχουμε τα Εστονικά, ή στη Δυτική Ευρώπη, τα Ιρλανδικά, τα Γκάιλικ. Όλα, όλες αυτές οι γλώσσες είναι μέλη του NPLD, είτε πλήρη είτε όχι, με στόχο να γνωρίσουν καλύτερα εμέν τους δε, να δουν τι πολιτικές εφαρμόζονται στην Ευρώπη και επίσης υπάρχει και συνεργασία με διάφορα όργανα όπως είναι η Κομισιόν ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης δραστηριοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δοθεί μεγαλύτερη προβολή στις διάφορες γλώσσες και να μπορούν να έχουν και βάρος και φωνή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το NPLD λοιπόν είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των λαών της Ευρώπης και των γλωσσών τους, για να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας. Αυτή οι δεσμοί είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμη, δύο σήμερα, που βλέπουμε να υπάρχει μια ανησυχητική διαίρεση, ένα χάζο μεταξύ βορρά και νότου στην Ευρώπη. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές το εξή. Το NPLD δεν περιλαμβάνει γλωσσικές κοινότητες που είναι νοσταλγοί του παρελθόντος και που το μόνο τους ε, ενδιαφέρον είναι ε, ένα εθνικιστικό παρελθόν να αναβιώσει. Σε καμία περίπτωση εμείς θέλουμε να σχετίσουμε μεταξύ τους τις γλώσσες που αντιπροσωπεύουν τις ρίζες των παρελθόν ε, των ευρωπαϊκών κοινωνιών και επικεντρώνουμε το έργο μας σε θεματικούς τομείς, την οικονομία, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, το ρόλο που έχουν όλες οι γλώσσες αυτές τις πτυχές, κινητικότητα, μετανάστευση ή οι γλώσσες ως παράγοντας κοινωνικού δυναμικού, κοινωνικής δυναμικής. Επίσης προσπαθούμε να προωθήσουμε και ένα οδικό χάρτη για την γλωσσική πολυμορφία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διάφορες γλωσσικές κοινότητες. Ό,τι αφορά την ε, διασύνδεση γλωσσών και οικονομίας, έχουμε αναθέσει στον καθηγητή Φρανσουά Γκρά από τη Γενέβη. Ε, τον θέσαμε λοιπόν μια μελέτη να μελετήσει ε, τη θέση που έχουν οι γλώσσες μεσαίου ή μικρού μεγέθους στην οικονομία. Τα συμπεράσματα της έκθεσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για τη σχέση μεταξύ των γλωσσών και την αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας για την Ευρώπη. Δεν χωρί αμφιβολία ως προς το ότι οι γεμονικές γλώσσες όπως τα γαλλικά, τα αγγλικά ή τα ισπανικά επηρεάζουν, η γλώσσα δηλαδή αυτών των γλωσσών επηρεάζει την κατάκτηση ενός υψηλοαξιώματος. Επίσης, στην έκθεση γίνεται λόγος για την ανάγκη προώθησης των τοπικών γλωσσών, ακριβώς για να προωθηθεί η ζωτικότητα της τοπικής οικονομίας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε σημερινούς καιρούς που βιώνουμε. Μια άλλη ε, σκέψη που βλέπουμε να αναπτύσσεται στην έκθεση είναι πώς επηρεάζει η γλωσσική πολυμορφία και η πολυγλωσσία τη δημιουργικότητα, την καινοτομία. Δεν θα πρέπει να ξεχάμε ότι όλοι όσοι μιλούν μια μειονοτική γλώσσα μιλούν και μια γλώσσα την οποία μιλεί η πλειονότητα της χώρας. Ας πούμε, ένας ε, που μιλάει ε, κορσικά δεν, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλάει και γαλλικά ή ένας καταλανός που μιλάει καταλανικά δεν υπάρχει περίπτωση να μιλάει ισπανικά. Για να σας δώσω δύο παραδείγματα. Όλοι μας σχεδόν είμαστε το λιγότερο δίκλωση για να μην πω πολύγλωση. Αν τώρα δούμε τη σχέση μεταξύ κινητικότητας μετανάστευσης και γλωσσών, το NPLD επίσης ανέθεσε μία μελέτη για το θέμα αυτό, για οικονομικούς λόγους, ε, για αγάπη, για άλλους ε, λόγους. Οι κάτοικοι, δεν μιλάω αυτούς που έχουν διαβατήριο, οι κάτοικοι μιας χώρας είναι όλο και πιο κινητικοί. Έχουμε παραδείγματο έναν Καταλανό που γεννήθηκε στην Καταλωνία, μιλάει Ισπανικά, Καταλανικά και έρχεται στην ε, στο Βέλγιο, για να βρει ε, θέσει εργασία και γνωρίζει όχι μόνο, δεν αποκτά μόνο μια δουλειά, αλλά ε, γνωρίζει την αγάπη. Παντρεύεται, αποκτά δύο παιδιά. Τα παιδιά του μιλάνε Ολλανδικά, Γαλλικά, μιλάνε Αγγλικά, μαθαίνουν Αγγλικά στο σχολείο. Πέντε γλώσσε δηλαδή. Ή ένα Μαροκινό που μιλάει μαζί ή αραβικά έρχεται να ζήσει παραδείγματο χάρη στη χώρα των Βάσκων και μαζί με τις δύο αυτές γλώσσες τα παιδιά του θα μάθουν και ισπανικά και βασκικά. Είναι Ευρωπαίοι πολίτες αυτοί. Ε, και οι Ευρωπαίοι πολίτες γενικά χαρακτηρίζονται από ε, αυτή την πολυμορφία, την γλωσσική. Αν υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση, η διατήρηση όλων αυτών των γλώσσεων δεν θα είναι πρόβλημα για τι μελλοντικέ γενιέ, αλλά θα ε, συνιστά σημαντική αξία και για τη γεωγραφική κινητικότητα, αλλά και την κοινωνική κινητικότητα των ατόμων. Με άλλα λόγια, η πολυγλωσία, αυτή η προσωπική και κοινωνική πολυγλωσία είναι ένας, από, είναι ε, ένας πλούτος για την Ευρώπη. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι μια μονόγλωση Ήπειρος ε, θα εξοικονομούσε κόστος και θα ήταν πιο αποτελεσματικό. Αυτό δεν ισχύει. Εμείς θέλουμε να αναλύσουμε τα ωφέλη της πολυγλωσσίας για την οικονομία, την αγορά εργασίας, την κοινωνική συνοχή, την κινητικότητα Γι' αυτό και επί Ιρλανδική Προεδρία θα δρομολογήσουμε τον οδικό χάρτη για την γλωσσική πολυμορφία. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία στηρίζει ο Ευρωβουλευτή που είναι μπροστά μου, ο κύριο Φρανσουά Αλφονσί, η κυρία Κιγκαγκάλ από το Intergroup, ε, το σχετικό. Όλοι σας είστε προσκεκλημένοι στην εκδήλωση αυτή. 11 Απριλίου θα λάβει χώρα στην Ιρλανδική Πρεσβεία εδώ στις Βρυξέλλες και θα έχει ως βασικό στόχο να εξασφαλίσει το ότι η Ευρώπη δεν θα ξεχάσει το μεγάλο δυναμικό που αντιπροσωπεύουν όλες οι γλώσσες. Όλες, τονίζω αυτή τη λέξη. Συχνά Κατηγορείται για δημοκρατικό έλλειμμα η Ευρώπη και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ποιότητα μιας δημοκρατίας μετράται και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις μειονότητές της. Η γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης είναι μια δυναμική και μεταλλασσόμενη πραγματικότητα. Το NPLD πιστεύει, εργάζεται ω προς, το σκοπό, ως το σκοπό την επίτευξη του στόχου της αμοιβαία ε, ε, και για όλους εποφελούς ε, ένταξη όλων των γλωσσών στην Ευρώπη. Πρέπει να ατενίσουμε θετικά όλες τις γλώσσες, να τις αντιμετωπίσουμε ως αξία, ως περιουσιακό στοιχείο, το οποίο όλοι οι λαοί της Ευρώπης θα πρέπει να έχουν ως κοινό. Εργαζόμαστε για να πετύχουμε ισότιμη πολυγλωσία στην Ευρώπη, για το σεβασμό της διαφορετικότητας και η πολυγλωσία θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των γλωσσικών κοινωνιών και κοινοτήτων. Θα είναι και ένα μέσο, ένα όχημα διαλόγου μεταξύ των διαφόρων κοινωνιών. Βέβαια το έργο μα. δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε την στήριξή σα, τη στήριξη των Ευρωβουλευτών, τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των γλωσσικών κοινοτήτων για να μπορέσουμε να πετύχουμε του κοινού μα στόχου. Μόνο με κοινή δουλειά όλε οι ευρωπαϊκέ γλώσσε θα μπορούν να ε, μιλούν με μία φωνή. Ευχαριστώ. head Τώρα λοιπόν έχουμε τον ε, κύριο Chris Jones, τον επικεφαλής ε, του οργανισμού αυτού. Εσείς έχετε PowerPoint. Πολύ ωραία. Good morning. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω ενώπιον σας σήμερα και ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη αυτή η παρουσίαση PowerPoint. Τις περασμένες εβδομάδες συνέτασα την έκθεση για τις ε, από, ε, από εξαφάνιση απειλούμενες γλώσσες και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, την εμπειρία που απέκτησα εργαζόμενο σε αυτό το τομέα και επίσης να σας δώσω κάποιες εξηγήσει σε σχέση με την ε, σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη ως προς αυτές τις γλώσσες. Εξυπακούεται ότι οι τρεις προλαλήσαντες ήδη σας έδωσαν πολλές πληροφορίες και ε, ε, έκαναν κάποιες παρατηρήσεις και τις ενέγραψαν σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Τώρα, ποια είναι η σχέση αυτών των γλωσσών με τις ε, γλώσσες μειονοτήτων. Δεν υπάρχει πραγματικός ε, ορισμός για την απειλούμενη γλώσσα στην UNESCO. Έχουμε αυτές τις κατηγορίες ε, που προαναφέρθηκαν, αλλά σε σχέση με το τι εστί απειλούμενη γλώσσα ανακύπτουν διάφορες δυσκολίες. Υποθέτω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις γλώσσες για να δώσουμε έναν ορισμό. Υπάρχει μια ad ομάδα που συστάθηκε από την UNESCO η οποία ισχυρίζεται ότι απειλείται η γλώσσα όταν οι χρήστες της σταματούν να την ε, ομιλούν, να τη χρησιμοποιούν. Όμως οι γλώσσες που δεν θεωρούνται εθνικές, οι περισσότερες γλώσσες που δεν είναι εθνικές εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Άρα όλες είναι απειλούμενες. Ε, ας προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τη γλώσσα, τις απειλούμενες γλώσσες, ε, αλλά σίγουρα χρειάζεται ε, περισσότερη δουλειά, διότι ε, θα πρέπει αυτός ο ορισμός να καλύπτει αυτές τις γλώσσες τώρα και μελλοντικά. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι έχουμε και το ψήφισμα του Νοεμβρίου 2008 του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, όπου ε, αναφερόταν ε, τι σημαίνουν οι γλώσσες στην Ευρώπη, δηλαδή είναι κοινό κληροδότημα, ένας πλούτος και ίσως και μια πρόκληση Νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί συνιστούν πλεονέκτημα αυτές οι γλώσσες για την Ευρώπη. Επίσης συνιστούν μια δέσμευση από πλευράς της Ευρώπης. Ποια είναι η αξία μιας γλώσσας αναρωτιέται κανείς ε, τι αξίζουν αυτές οι γλώσσες, γιατί πρέπει να τις κρατήσουμε, γιατί πρέπει να ε, ε, μπορούν κάποιοι να μιλούν ουελικά. Θα ήταν απλούστερα τα πράγματα αν δεν είχαμε τόσες γλώσσες. Λοιπόν, ποια είναι η αξία των γλωσσών ως προς τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή για να υπάρχει ένας καλύτερος οικονομικός ρυθμός, πιο ρηξικέλευτος αν θέλετε, συνειδητοποιούμε ότι όσοι μιλούν πάνω από μία γλώσσα ε, είναι πιο ε, ενιολογικά δημιουργικοί σε σχέση με αυτούς που μιλούν μόνο μία γλώσσα. Αυτό μας δείχνει η έρευνα ως προς τη δημιουργικότητα των ανθρώπων και τις ευαισθησίες που έχουν σε επικοινωνιακό επίπεδο. Ε, πολύ σημαντική πτυχή επίσης. Πέραν αυτών υπάρχει και μια πτυχή που εντοπίζεται στα ΜΜΕ, στις δημιουργικές οικαστικές τέχνες. Πρόκειται για μια ε, διαφορετική γνωστική ικανότητα που έχουν όσοι ομιλούν περισσότερες γλώσσες. Έγινε μία παραγουσία σε σχέση με το πόσες γλώσσες ε, ε τέτοιες υπάρχουν στον κόσμο. Ανάμεσα στις 6 και 7 χιλιάδες υπολογίζονται. 96% των γλωσσών σε παγκόσμιο επίπεδο μιλούνται από μόνο το 3% του παγκοσμίου πληθυσμού. Οπότε οι γλώσσες μειονοτήτων και οι απειλούμενες γλώσσες εγγράφονται στο ίδιο πλαίσιο τρόπον την... Οι περισσότεροι άνθρωποι ομιλούν πλειοψηφικές ε, γλώσσες. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στι δύο κατηγορίες από αυτή την πλευρά. Ας δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Πόσες γλώσσες μιλούνται στην Ευρώπη. Μόνο 3% των γλωσσών... Ε, των, Ηθαγενών ομιλούνται ε, από, στην Ευρώπη και ε, δεν ε, θα μπορέσουμε ε, λοιπόν στην Ευρώπη να έχουμε την ίδια προσέγγιση όπως σε άλλα μέρη του κόσμου όπου το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο. Τώρα, το πρόβλημα του ορισμού είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Όταν μιλάμε για την ύπεθρο και ε, περιοχές που οικονομικός πώς είναι σε δυσμενέστερη θέση, δεν αποτιμούνται στη σωστή αξία τους οι γλώσσες, δεν έχουν το καθεστώς που τους αναλογεί και Άρα παρακολύεται η διαγενειακή μετάδοση των γλωσσών. Ως προς εργασίες ε, της UNESCO θα δείτε ότι υπάρχει μια σειρά κριτηρίων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποφασίσουμε αν απειλείται μια συγκεκριμένη γλώσσα ε, και τι ακριβώς δεν συμβαίνει σε αυτή τη γλωσσική κοινότητα. Ε, δεν υπάρχει ακριβώς αυτή η διαγενειακή μετάδοση. Είναι μικρός αριθμός ε, των ομιλητών, μικρός αριθμός των τομέων όπου χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα. Τέτοια κριτήρια χρησιμοποιούνται για να καταλήξουμε σε έναν ορισμό αυτών των γλωσσών. Ω προ τι επίσημε γλώσσες, γλώσσες εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι ε, ε, γλώσσε ε, περιφερειακού χαρακτήρα. Υπάρχουν, και οι γλώσσες οι ή μη επίσημες, οι λεγόμενες, Όλες αυτές οι γλώσσες χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά καμία τους δεν έχει ένα επίσημο καθεστώς. Πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια διαφορετική περιγραφή αυτών των γλωσσών. Όποιον όρο και αν επιλέξουμε για να τις περιγράψουμε, συνειδητοποιούμε ότι κάποιες γλώσσες υπάρχουν μόνο ε, σε ένα κράτος. Αυτόχθονες γλώσσες ονομάζονται αυτές. Έχουμε και άλλη κατηγορία Πέρα από τις αυτόχθονες έχουμε και τις διασυνοριακές γλώσσες ε, οι οποίες δεν είναι ε, ε, οι πλειοψηφικές σε πάνω από μία χώρα. Στα βασικά παραδείγματο χάρη στην Ισπανία και τα βασικά στη Γαλλία. Στη συνέχεια, διασυνοριακές γλώσσες, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, είναι πολύ άριθμες αυτές οι διασυνοριακές. Επίσης, μη εδαφικές γλώσσες, όπως η διάλεκτος των Ρωμά. Ε, ε, τέτοια ε, προβλήματα αντιμετωπίζουμε όταν προσπαθούμε να ταξινομήσουμε όλες αυτές τις γλώσσες. για τον Άτλαντα τώρα δίνει, προσδίδει μία δομή στον τρόπο ταξινόμησης των απειλούμενων γλωσσών. Όμως αν δείτε το επίπεδο προστασίας που προσφέρει αυτή η χάρτα, βλέπουμε ότι οι απειλούμενες γλώσσες τείνουν να υπάγονται στο, στο πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα είναι αυτό όπου τα κράτη-μέλη με κάποια λεπτομέρεια περιγράφουν τι είδους προστασία προσφέρουν για αυτές τις ε, χώρες. Οι απειλούμενες γλώσσες ε, υπάγονται όμως αυτήν την ε, πρώτη κατηγορία όπου δεν παράσχεται καμία προστασία από τα κράτη-μέλη. Ας προχωρήσω τώρα στο ζήτημα της χρηματοδότησης. Βλέπουμε και πάλι ότι ο μόνος γνώμονος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι αυτός που σχετίζεται με τις μειονεκτικές γλώσσες. Υπήρχε μια γραμμή χρηματοδότησης από το 83 και μετά και μέχρι το 1998 φτάσαμε τα 84 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων. Όμως αυτό ε, θεωρήθη έκνομο στα τέλη της ε, δεκαετίας του 90 και έπαυσε αυτή η χρηματοδοτική δραστηριότητα και οι τελευταίες πληροφορίες είναι από την Επιτροπή των Περιφερειών το 2011. Αναφέρεται σε ένα ψήφισμα ότι η συγκεκριμένη γλωσσική πολιτική για τις ε, μειονεκτικέ γλωσσικές κοινότητες ε, δεν ε, χαίρει επαρκού χρηματοδότηση Αυτά για τη χρηματοδότηση και την προστασία των γλωσσών για να υλοποιηθούν προγράμματα ή να αυτοσυντηρηθούν αυτέ οι γλώσσε. Σε αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες και έγγραφα πολιτικής για την ε, υποστήριξη της γλωσσικής ε, πολυμορφίας και της πολυγλωσσίας. Ε, δεν θα διατρέξω αυτό το μακρύτατο κατάλογο δράσεων τα τελευταία χρόνια προς υποστήριξη της πολυγλωσσίας. Έγινε και μια δημόσια συζήτηση σε σχέση με τον τρόπο που πρέπει να προστατεύονται αυτές οι γλώσσες. Χρειαζόμαστε οργανισμό, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά δίκτυα. Το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτεινε προς τα δίκτυα και υπάρχουν κάποια δίκτυα που έχουν συσταθεί όμως δεν ε, είναι επαρκής η χρηματοδότησή τους. Κάποια κράτη-μέλη επίσης ε, ε, έχουν ε, λίγο εξελιγμένες πολιτικές για να χειριστούν αυτό το θέμα των μειοψηφικών γλωσσών στην επικράτειά τους. Υπάρχει κείμενη νομοθεσία ενίοτε, χρηματοδοτούνται προγράμματα και κάποια κράτη-μέλη, αλλά όχι πολλά, προστατεύουν τις απειλούμενες γλώσσες. Εν γενή, οι καλύτερες στρατηγικέ είναι για τις πλειοψηφικές γλώσσες. Για τις απειλούμενες γλώσσες δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ε, η και μεγαλύτερη ευκαιρία των απειλουμένων γλωσσών είναι η τεχνολογία και τα κοινωνικά δίκτυα. Ε, αν προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε τη δράση μα για το μέλλον, τα κοινωνικά μέσα μαζική ενημέρωση είναι ένα τρόπο να υποστηρίξουμε αυτέ τι γλώσσε με μικρή υποδομή. Βεβαίω, ε, οι ομιλητέ και χρήστε αυτών των γλωσσών πρέπει να κρίνουν ε, οι ίδιοι ότι είναι αρκετά σημαντική η γλώσσα του για να στέλνουν μηνύματα tweet ε, σε αυτή τη γλώσσα, παραδείγματο χάρη. Όταν μιλάμε για αυτέ τι γλώσσε, συνειδητοποιούμε ότι όταν χάνεται μία γλώσσα, χάνεται ΣΑΗ, ε, διαπαντός. Ε, βλέποντας λοιπόν τις απελούμενες γλώσσες, αν θέλουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι γλώσσες, ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε υποστήριξη για αυτές. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει και το ζήτημα της επικουρικότητας. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως τίθεται και ένα ζήτημα για τις απελούμενες γλώσσες. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται για εγκάρσια ευθύνη που καλύπτει ε, για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία οφείλει να προστατεύσει ε, την ε, γλωσσική της μορφία και απαντώνται τέτοιες συστάσεις σε διάφορα νομοθετήματα. Ποιος είναι όμως ο ορισμός της επιτυχημένης δράσης σε αυτό το τομέα. Ε, κάποιος θα αρχίσει να μιλάει ε, στη, το Σάββατο το βράδυ ε, στο δρόμο μια απειλούμενη γλώσσα. Πώς ένας 20χρονος μπορεί να αρχίσει να μιλάει αυτήν την γλώσσα. Αυτό συνιστά ευκαιρία και πρόκληση για τα κράτη-μέλη. Βλέποντας όμως την πραγματική εικόνα της Ευρώπης, χρειάζεται δημόσιος διάλογος. Με ποιο τρόπο όντως μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτές τις απειλούμενες γλώσσες και να εξασφαλίσουμε ότι η γλωσσική ομοσπονδία της Ευρώπης ε, θα διασφαλιστεί. Σας ευχαριστώ, εμείς σας ευχαριστούμε. Έχουμε τώρα ένα πακτολό πληροφοριών και συστάσεων. Δεν είναι εύκολο να δοθεί η σωστή απάντηση, διότι ε, όπως σωστά είπατε υπάρχει η δαμόκλειος πάθη της επικουρικότητας ε, που κρέμεται πάνω από, πάνω από μας Σίγουρα καταβάλουμε προσπάθειες, αλλά δεν είναι ότι έχουμε ε, σεντούκια με λεφτά έτοιμα που μας περιμένουν. Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την παιδεία στα πλαίσια της δημιουργικής Ευρώπης. Ε, φυσικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, τέτοιες δράσεις, αλλά το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να, ευαισθητο... να κάνουμε εξτρατείες ευαισθητοποίησης των περιφερειών ε, για να δράσουν από μόνες του γιατί δεν έχουμε επαρκή κονδύλια. Ευχαριστούμε πάντω για όλες τις πληροφορίες. Και τώρα ε, θα αρχίσουμε με τις έρωτα απαντήσεις. Φίθια Σαντιάγκο, ε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αλφονσί που είναι ο συγγητής της σημαντικής αυτής έκθεσης και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ομιλητές που μας ε, παρουσίασαν αυτό το θέμα σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνώ με την άποψη ότι οι μειονοτικές γλώσσες πρέπει να την χάνουν προστασίας. Σίγουρα έγινε λόγος για πολλούς ορισμούς. Είναι δύσκολο να ορίσουμε αυτές τις ε, γλώσσες. Έχουμε τις γλώσσες στις οποίες κάποιος ε, προσεύχεται, ε, ονειρεύεται. Και ο Κάλλος Σαπέτς χρησιμοποιούσε μια... είχε πέντε γλώσσες που μιλούσε και για κάθε περίσταση διαφορετική χρησιμοποιούσε ανάλογα και μια άλλη γλώσσα. Εμένα αυτό το οποίο λίγο με προβληματίζει ο τίτλος της έκθεσης Εγώ νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα δύο κομμάτια αυτής της έκθεσης. Δηλαδή, άλλο οι ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και άλλο η γλωσσική πολυμορφία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους τα δύο αυτά. Γι' αυτό θα ήθελα να μας εξηγήσετε ακριβώς, κύριε Αλφονζή, πού θα επικεντρωθείτε στην έκθεσή σας. Θα επικεντρωθείτε στις ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση ή και στη γλωσσική πολυμορφία. Η πρόεδρος μας, η Ντόρι Πακ, είπε ότι θα δεχθείτε μόνο τροπολογίες οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα τις γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση. Αλλιώς δεν θα δεχθείτε, είπατε, καμία τροπολογία, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο με εκπλήσει λίγο είναι το έγγραφο που μας μοιράσατε για τις γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση. Συγγνώμη που θα μιλήσω για την Ισπανία, αλλά λέτε ότι τα βασικά απειλούνται με εξαφάνιση. Μα είναι μια προστατευμένη γλώσσα, είναι επίσημη γλώσσα στη χώρα των Βάσκων και στην περιοχή της Ναβάρα, διδάσκεται στα σχολεία. Ενώ το αρανές, μειονοτική γλώσσα που μιλάτε στην κοιλάδα του Αράν, πάρα πολύ ωραία περιοχή βέβαια, εκεί είναι επίσημη, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο διαφορετική κατάσταση από μια γλώσσα στην άλλη, σε ό,τι αφορά δηλαδή τον κίνδυνο εξαφάνισης. Σε ένα άλλο τώρα έγγραφο στα Ιταλικά, το έχω μπροστά μου, φαντάζομαι το έχουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, εκεί γίνεται λόγος για τις διάφορε μονοτικέ γλώσσες στα διάφορα κράτη. Σε ό,τι αφορά τα καταλανικά, λέει ότι μιλείτε, ομιλείτε μόνο στην Ισπανία. Δεν ισχύει αυτό και στη Σαρδινία ομιλείται και φυσικά και στην Γαλλία. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που είπε ο κύριο Θεράνου, είναι σημαντικό όχι μόνο το να ομιλείτε μια γλώσσα, αλλά και η ποιότητα. Πώς δηλαδή ομιλείτε μια γλώσσα. Είπατε Κύριε Αλφόνσο, δεν ξέρετε κανέναν ε, στην ε, Ισπανία, ε, στη, μάλλον στην Καταλωνία, που δεν μιλάει Ισπανικά. Ναι, αλλά ξέρω πολλούς Καταλανούς εγώ στην ε, Καταλωνία που μιλάνε φρικτά Ισπανικά. Άρα δεν αρκεί να μιλάει κανείς, το θέμα να ξέρει και τι λέει. Να έχει μια ποιότητα η γλώσσα δηλαδή. Επικοδομητική πάντως θα είναι η έκθεση γιατί τα διά, οι διάφορες γλώσσες είναι ε, κομμάτι της κληρονομιάς της ευρωπαϊκής. Και όχι μόνο οι γλώσσες. Μειονοτικά ε, αθλήματα, μειονοτικά σπορ σε, κάποιους, ε, σε κάποιες περιοχές ασκούνται. Και θα έχουμε στο ΕΛΚ και μία ημερίδα για την προστασία αυτών των μειονοτικών αθλημάτων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία κάμεραβέρτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ επίσης και για τις ε, ομιλίες που ακούσαμε. Εκείνο που κατάλαβα και νομίζω αυτό θέλω να το προτείνω και στον συνάδελφο Αλφόνζη, είναι ότι θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τον ορισμό ε, και τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε γλώσσα απειλούμενη από εξαφάνιση και γλώσσα μειονότητα. Ε, κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ή αν είναι τελικά το ίδιο. Εμείς στο γραφείο μου ε, βρήκαμε μία μελέτη όπου γίνεται λόγος για την εξαφάνιση γλωσσών λόγω της ψηφιοποίηση. Και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή περίπου 200 γλωσσολόγοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ολόκληρο τον κόσμο εντόπισαν ή ερεύνησαν 30 ευρωπαϊκές γλώσσες και αυτές που ξέρουμε, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, εστονικά, λετονικά, όλες αυτές τις γλώσσες, εν πάση περιπτώσει, και είδαν πως ε, στηρίζονται τεχνολογικά αυτές οι γλώσσες. Δηλαδή, αν ε, στηρίζονται από μεταφραστικά προγράμματα, αν υπάρχουν ε, προγράμματα ορθογραφίας ε, στον υπολογιστή, στο λογισμικό που να βοηθούν. Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι 21 από αυτές τις 30 σε όλους μας γνωστές γλώσσες απειλούνται και μάλιστα ουσιαστικά λόγω της ψηφιοποίησης. Αυτό λοιπόν το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι κάτι που νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε κάποιες γλώσσες που τις θέλουμε. Μας αρέσουν πολύ τα γερμανικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, λετονικά, εστονικά και οτιδήποτε άλλο. Οι γλώσσες αυτές να μην εξαφανιστούν και λόγω της διάδοσης ε, της τεχνολογίας. Απλά και μόνο διότι δεν τα στηρίζονται από λογισμικά. Και εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, ε, εντείνεται αυτή η τάση να μιλάνε όλοι μία γλώσσα που σημαίνει τελικά αγγλικά. Εντυρωτήθηκα λοιπόν το εξή κατά πόσον στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε ε, και να συμφωνήσουμε ως προς το ότι ορισμένες γλώσσες απειλούνται. Θυμάμαι τη συζήτηση που κάναμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπεται αυτό να συζητηθεί σήμερα και στην διάρκεια της συνεδρίασης των συντονιστών πέρυσι, στο πλαίσιο μιας μεγάλης πρωτοβουλίας, καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέπει τις διαβουλεύσεις σε όλες τις ε, ευρωπαϊκές γλώσσες, ε, να επιτρέπει την αλληλογραφία σε όλες αυτές τις γλώσσες. Έκτοτε όμως η Κομισιόν αρνείται στεναρά και λέει ότι εμείς ε, διαβουλευόμεθα μόνο σε γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά. Αυτό λοιπόν εγώ το ορίζω ως ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν και εμείς εδώ στην Ευρώπη λέμε μόνοι μας ότι επιτρέπουμε μόνο τρεις γλώσσες ε, και όποιος άλλος ε, θέλει να απευθυνθεί στην Κομισιόν σε άλλη γλώσσα να είναι σίγουρος ότι δεν θα μεταφραστεί και να είναι σίγουρος ότι δεν θα πάρει την απάντηση στη γλώσσα του. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα θα συζητήσουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα αυτό. Ξέρουμε βέβαια ότι έχει επιληφθεί του θέματος και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής. Για μας ε, είναι σημαντικό αυτή η πολυγλωσία ε, που υπάρχει στην Ευρώπη να προστατευτεί. Και για να γίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική μας και δεν ισχύει μόνο αυτό για το Κοινοβούλιο αλλά σε όλους τους ε, ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όλες οι γλώσσες είναι ισότιμες και ως τέτοιες αντιμετωπίζονται είτε από το Κοινοβούλιο είτε από την Κομισιόν είτε από το Συμβούλιο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε και θα μου επιτρέψετε ε, και να κάνω και μία ερώτηση προς τους εμπειρογνώμονές μας. Τι μπορούμε να κάνουμε ως Ένωση, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στηρίξουμε και όχι μόνο με κονδύλια, το είπε και η Πρόεδρος, δεν έχουμε πάρα πολλά κονδύλια. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε έτσι ώστε πέρα από την οικονομική υποστήριξη να μπορέσουμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε ε, πραγματικά να διατηρηθεί η πολυγλωσία στην Ευρώπη σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Ε, ευχαριστούμε. Κέλλη παρακαλώ. Ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες για τη συμβολή τους. Είμαι Ιρλανδός και εκεί έχουμε τα Ιρλανδικά, φυσικά, τη μειονεκτική γλώσσα και έχω την τιμή να τα ομιλώ. Ε, και οι έχουν, παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την μετάφραση τέτοιων γλωσσών σε θεσμικά όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για όλες τις μειονεκτικές γλώσσες, αυτές που θεωρούνται μειονεκτικές. Το εκτιμούμε ιδιαίτερως. Είναι περιορισμένα τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για την προώθηση αυτών των ε, γλωσσών. Ε, Φερρυπίν, ε, μπορώ να μιλήσω εδώ Ιρλανδικά και θα μεταφραστώ. Ε, είναι κατανοητό το ότι είναι περιορισμένα τα κονδύλια γιατί δεν μπορούν να δεν μπορούμε να διαθέσουμε τελείωτα κονδύλια. Ε, γι' αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, ε, και τις τεχνολογίες, ώστε οι νέοι να μιλούν περισσότερο αυτές τις γλώσσες, αλλά ε, είναι περιορισμένη η δράση μα, διότι παραδείγματο χάρη την ιστοσελίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ θα, δεν θα την ε, ποτέ θα μεταφραστεί στα Ιρλανδικά. Ε, ούτε και κάποια κείμενα νομοθετικά, όπω η συνθήκη τη ε, Λισαβόνα και ποιο θα πάει να την ψάξει και όλα στη μεταφρασμένη εκδοχή και ακόμη και αν μεταφραστεί. Οπότε πρέπει να εστιάσουμε στους τομείς όπου θα είναι πιο αποδοτική η δράση μας. Ε, πρέπει να μιλούνται. Προφορική χρήση των γλωσσών. Αυτό, αυτή είναι η σημαντικότερη διάσταση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έπρεπε μέσα από τα κοινωνικά ΜΜΕ να επιδιώξουμε αυξημένη προφορική χρήση των γλωσσών. Ε, κάτι τώρα ε, ιδιαίτερα θετικό που ακούσαμε ε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος ακούστηκε ότι υπάρχει οικονομική επιχειρηματολογία υπέρ των μειονεκτικών γλωσσών παρόλα αυτά ε, στατιστικά δεδομένα βάσει των οποίων 97% του παγκοσμίου πληθυσμού μιλούν 4% του αριθμού των γλωσσών που υπάρχουν στην Ιφίλιο. Ε, όμως ε, μπορούμε να πούμε, να γενικεύσουμε και να στρογγυλέψουμε αυτά τα ποσά και να πούμε, ορίστε, το 100% μιλούν μόνο το 4% των γλωσσών και λύνεται το πρόβλημα. Όμως πώς μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οικονομικός πώς είναι επικερδής η χρήση αυτών των ε, μειονεκτικών γλωσσών. Αυτό διαπιστώνω και στη χώρα μου. Ε, όσοι μιλούν μεγάλες γλώσσες όπως ε, τα αγγλικά ή τα γαλλικά είναι πιο απασχολήσιμοι σε εισαγωγικά σε σχέση με τους μονόγλωσσους. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν να προσποιούμαστε. Η αξία μιας γλώσσας, κάτι που μας απασχόλησε νωρίτερα, είναι κομμάτι της κουλτούρας και είναι αυτός σκοπός η συντήρηση μιας τέτοιας γλώσσας. Βεβαίως χρειάζονται χρήματα για την προώθηση αυτών, αλλά δεν μπορώ να ε, καταλάβω πώς μπορείτε να το πείτε. Εγώ δεν μπορώ να πάω στην, ε, στην Ιρλανδία και να τους πω ότι αν, το, αν προωθήσετε τα Ιρλανδικά θα αυξηθεί κατά τόσο το ΑΕΠ της χώρας και θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερες λεπτό σε σχέση με αυτό. Εγώ θέλω να προστατευθούν, να διατηρηθούν οι γλώσσες και κυρίως να ε, δημιουργήσουμε κινήτρα τόσο ώστε να χρησιμοποιούν οι νέοι αυτές τις γλώσσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Τόρκες τώρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον κορσικανό συνάδελφό μας, τον κύριο Αλφόνση, να έχει επιληθεί του ζητήματος ε, των ε, απειλημένων γλωσσών. Είμαι ο σκιώδης συζητητής του ΕΛΚΕ για αυτό το ζήτημα και θα ήθελα απευθείας να δηλώσω ότι ε, θα συνεργαστώ μαζί του ως ε, ε, ε βουλευτής που ανήκω στην ε, κοινότητα Ρωμά ταυτόχρονα. Συγγνώμη που έρχομαι από την Ουγγαρία και από τη Ρουμανία και στη Ρουμανία ε, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε ε, ουγγρικά στο σχολείο ούτε καν στο διάλειμμα δεν επιτρεπόταν ε, στην αυλή, στο προάβλιο δεν ε, είχαμε το δικαίωμα να μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα διότι θεωρείται η γλώσσα του διαβόλου. Ε, και αν κάποιος ε, ήθελε στη Ρουμανική Βουλή να μιλήσει ουγγρικά θα δημιουργούσε αυτό ένα πελώριο σκάνδαλο. Ε, αντίθετα εδώ με φυσιολογικό τρόπο μπορούμε να μιλήσουμε όποια γλώσσα θέλουμε και με ικανοποιεί ιδιαίτερα αυτό το γεγονός. Μιλώντας για το οικονομικό δυναμικό των γλωσσών είναι κατά τι τεχνητό αυτό το επιχείρημα. Ακόμη και αν οι μικρές απειλούμενες γλώσσες δεν έχουν ε, ε, ουσιαστική οικονομική αξία, θα πρέπει να προστατευτούν διότι έχουν ε, μια διαφορετική αξία πέραν της οικονομικής. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές. Γιατί να προστατεύουμε την βιοπικιλότητα και όχι την γλώσσοπικιλότητα. Γιατί ασχολούμαστε με όλο αυτό τον αριθμό των ε, ε, ειδών ε, υπό εξαφάνιση, αλλά όχι με τις από εξαφάνιση απειλούμενες γλώσσες. «700.000 Σουηδοί και Ούγγροι στην Τρανσιλβανία Σουάβοι και Σαξόνοι ε, ε, έφυγαν από την ε, Τρανσιλβανία και εξέλιψαν 700.000 άνθρωποι, χάθηκαν χωριά, εκκλησίες, σπίτια. Είναι μεγάλες οι απώλειες παρά τις προσπάθειες που έγιναν για την προστασία τους. Πριν από 100 χρόνια Υπήρχαν πολύ περισσότεροι Ούγγροι, λειτουργούσαν πολλές περισσότερες εκκλησίες και τώρα όταν επισκέπτομαι αυτά τα χωριά είναι θλιβερή εικόνα Από αυτή την άποψη δεν θα συμφωνήσω απολύτως με την κυρία Πακ που μας λέει ότι δεν πρέπει να μιλούνται μειοψηφικές γλώσσες. Εγώ πιστεύω ότι οι απειλούμενες γλώσσες και οι μειοψηφικές γλώσσες είναι αλληλένδετες, δεν είναι δύο διακριτές κατηγορίες διότι οι καταπιεζόμενες ε, μειοψηφικές γλώσσες εξορισμού απειλούνται ε, από εξαφάνιση. Δεν μιλάω για τα όγκρικα στην Ουγγαρία, δεν απειλούνται στην Ουγγαρία, αλλά απειλούνται σε τουλάχιστον έξι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εκλείψει αυτή η γλώσσα σε αυτά τα έξι κράτη-μέλη αν δεν κάνουμε κάτι γιατί υπάρχει καταπίεση ως προς τη χρήση των ουγγρικών ε, που και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από διάφορες χώρες. Ε, και έχουμε και τους Σουηβούς ε, και τους Γερμανούς. Υπάρχουν και άλλες γλώσσες δηλαδή που απειλούνται στην επικράτεια της Ρουμανίας. Δεν είναι μόνο τα Ουγγρικά. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε για τις μειοψηφικές κοινότητες και όχι μόνο για τις μειοψηφικές γλώσσες που απειλούνται. Εν κατακλείδη θα ήθελα να σας μεταφέρω κάτι που συζήτησα με την Αγέλα Φέσσερ νωρίτερα. Στην ε, Τρανσιλβανία πριν από 50 χρόνια 80% ε, των ε, αθλημάτων γινόντουσαν στα Ουγγρικά και ο 80% των αθλητών, παραδείγματος χάρη στην ε, Ρουμανία, ήταν Ούγγροι. Αυτή η, αλλάξη, αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν σήμερα και δεν έχω κάτι κατά των Ρουμάνων αθλητών. Είναι πάρα πολύ καλή. Απλώς ε, θέλω να καταδείξω ότι υπάρχει μια τάση να ε, ε, εκλείπουν από τον επίσημο ή από τον αθλητικό βίο οι Ούγγροι στη Ρουμανία. Αν παραδείγματο χάρη θέλω να κάνω μια αθλητική σταδιοδρομία σήμερα, θα πρέπει να ξεχάσω ε, την γλώσσα μου για να παίξω στην εθνική ομάδα. Πολλοί άλλαξαν και το όνομά τους, το επώνυμό τους, για να μην ακούγεται ουγγρικό, για να μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν στον χώρο του αθλητισμού. Η Γιολάντα Μπέλους, παραδείγματος χάρη είναι ένα παράδειγμα αυτής της τάσης. Είμαι υπέρ ε, ε, της ε, προστασίας ε, των νέων στην Τρανσιλβανία για να μπορέσουν να συνεχίσουν να μιλάνε τη γλώσσα τους διότι το διακύβευμα είναι η ζωή της μειονότητας. Ευχαριστούμε κύριε Τόρκες. Κοιτάξτε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα νέο πρόβλημα το οποίο όμως θα σας το παρουσιάσω από ιστορική σκοπιά. Δηλαδή όταν ε, ε, τα ε, κράτη-μέλη, τα νέα, προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως όταν υπήρχε η εποχή του σιδηρού παραπετάσματος, τότε την εποχή εκείνη είχαμε πολλές μειονότητες οι οποίες καταπνίγονται λόγω συγκεκριμένης, στοχευμένης πολιτικής. Αυτή ήταν μια πολύ στοχευμένη πολιτική, όπως σας είπα, και όπως θέλω επίσης να προσθέσω, έχω πάρα πολλούς ε, φίλους οι οποίοι ανήκουν σε μειονότητες οι οποίες ε, μετακινήθηκαν ε, στο εσωτερικό ενός κράτους ή μετακινήθηκαν σε άλλα κράτη. Άτομα τα οποία δεν, είχαν, δεν τους επιτρεπόταν πλέον να μιλάνε τη γλώσσα τους γιατί θα αντιμετώπιζαν τεράστια προβλήματα. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε το αντίθετο, βλέπουμε την επιστροφή στις ρίζες. Δηλαδή τώρα πλέον γίνεται λόγος ε, για την προστασία του πολιτισμού και η γλώσσα είναι το όχημα των ε, ε, παραδόσεων και της ιστορίας. Αυτό λοιπόν για μένα είναι πολύ σημαντική αξία για τις εθνικές μειονότητες. Για αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά σήμαινε μια ουσιαστική αλλαγή. Και θα πρέπει και να πούμε και το εξή. Ε, παίζουμε πολύ σημαντικό ρόλο γιατί είμαστε η μόνη επιτροπή που ασχολείται με την προστασία των υποξαφάνιση απειλούμενων γλωσσών. Πρέπει να πέσει φως ε, στην ε, ιστορία των γλωσσικών μειονοτήτων γιατί το να είναι κανείς Ευρωπαίος πολίτης αυτή είναι μια θέση που πρέπει κανείς να την υπερασπιστεί. Και νομίζω ότι από την Επιτροπή μας πρέπει να εκπέμψουμε ηχηρό μήνυμα για να επισημάνουμε ότι η πολυγλωσία είναι μία από τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, βεβαίως και έχουν διαφορετικές ηθαγένειες ε, αλλά είναι ε, Ευρωπαίοι πολίτες αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω τώρα το δεύτερο Κατά το παρελθόν, εγώ ε, μία, συνέταξα μία έκθεση για τον Ευρωπαϊκό ε, Κινηματογράφο και αυτή η έκθεση δική μου ε, είναι συνδεδεμένη με το γλωσσικό. Στην Ευρώπη βιώνουμε γλωσσική κατάτμιση και στην Ευρώπη έχουμε μεγάλη παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. Ο κινηματογράφος λοιπόν είναι ένα στοιχείο για να ε, προστατεύσει κανείς ε, τον πολιτισμό του, να τον ε, προβάλλει, να τον παρουσιάσει σε διάφορους ανθρώπους. 200.000 ταινίες έχουμε το χρόνο στην Ευρώπη, δηλαδή διπλάσιο αριθμό ταινιών από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ένας Ισπανός, ένας Λιθωνός Κοιτάξτε, εγώ λόγω των, της τεχνολογίας που υπάρχει σήμερα πλέον μπορεί κανείς να γυρίσει μία ταινία ε, και με χαμηλό κόστος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δαπανίσει κανείς ε, περιουσία ολόκληρη για μία ταινία. Για μένα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά και απλά παραδείγματα. Ο ρόλος της δικής μας της Επιτροπής είναι το μήνυμα να είναι σαφές και δεν πρέπει πούμε να ξεχνάμε τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Ε, το πρόβλημα της Ισπανίας, όπου οι Ισπανοί δεν ήθελαν να ε, κυριαρχήσουν τελικά τρεις μόνο γλώσσες, αλλά η όλη διαδικασία ήταν σταδιακή, σε βήματα. τελικά αν ε, περιστούν, αν δεχτούμε να περιστούν οι γλώσσε τρεις, κινδυνεύουμε στο μέλλον να περιστούν ακόμα περισσότερο και να επικρατήσει μόνο μία που θα είναι τα αγγλικά. Μακροπρόθεσμα, εφόσον στηρίζονται οι γλώσσες, νομίζω ότι ε, προκύπτουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα ανεξάρτητα από το κόστος ε, που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υποστηρίζω όλους όσους συνιστούν τη διατήρηση και την προστασία των ενωτικών γλωσσών ως αυτό σκοπό. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το ζήτημα αυτού της ευρωπαϊκής γλωσσικής πολυμορφίας, ή μάλλον τη ευρωπαϊκής πολυμορφίας θα πρέπει να εντάξουμε σε αυτήν και τη διάσταση της γλωσσικής πολυμορφίας. Και εκεί να δώσουμε έμφαση. Και φυσικά όποιοι συνεισφέρουν στη διατήρηση της ε, πολυμορφίας πρέπει να στηριχθούν από την Επιτροπή μας, γιατί η γλώσσα είναι συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης ταυτότητας. τον Αριστοτέλη τον Τσόμσκι, όλοι οι γλωσσολόγοι λένε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Μάλλον μπορεί να έχουν τεράστια διαφορά μεταξύ τους αυτά τα δύο άτομα, αυτοί οι δύο γλωσσολόγοι, αλλά συμφωνούν απόλυτα προς το ρόλο της γλώσσας. κυρία Σουίνμπερν, αναπληρώτρια, βουλευτή στην Επιτροπή, πολιτισμού μου ζήτησε να διατυπώσω κάποιε παρατηρήσει εξ τη. τη. Κύριε Σουίνμπερν, είναι Αλή. και είπατε ότι η Ουαλία είναι μια περιοχή ε, και μια γλώσσα τα ολικά που πρέπει να προστατεύονται, να προστατευθούν. Και κυρία Σουίνμπερν δεν θεωρεί ότι υπάρχει μεν πρόβλημα, δηλαδή ότι οι Ουαλοί δεν είναι υπερήφανοι για τη γλώσσα τους, απλά όλο και λιγότεροι την ομιλούν στη χώρα αυτή, στην περιοχή αυτή. Η ε, κυρία Σύνμπρεν, λοιπόν, θα επιθυμούσε την εντατικοποίηση οποιασδήποτε δράσης που θα ήταν και να στηρίξει την ενολογογλώσσα αλλά και άλλες ε, γλώσσες σχετικές. Τονίζει επίσης την τεχνολογική πρόοδο που θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο, ένα πρόσθετο εργαλείο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει για να υποστηρίξουμε τις ε, γλώσσες που κινδυνεύουν να ξεχαστούν όπως είπε ο κ. Ε, η τελευταία παρέμβαση ήταν ίσως και πιο ενδιαφέρουσα. Κατ' εμέ τουλάχιστον. Η κυρία Σουίνμπερν επίσης θέλει να χαιρετήσει όλους τους ε, ομιλητές. Ακούσαμε κάποια σοκαριστικά στοιχεία. και αυτό ότι ε, το 90 περίπου τις 197% μιλάνε 4% των γλωσσών ήταν ένα στοιχείο Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στους εμπειρογνώμονες ε, για να απαντήσουν. Ε, έχουν στο χρόνο τους ε, κατά το μέγιστο 5 λεπτά και θα ήθελα πρώτα απ' όλους να δώσω το λόγο στον κύριο Jones, αν βέβαια το επιθυμεί. Εσείς θα μιλήσετε μετά αφού μιλήσουν οι εμπειρογνώμονες. Ο κύριο Jones. Κύριε Jones, θέλετε να λάβετε το λόγο. Θα μπορούσα να κάνω κάποια σχόλια για τις παρατηρήσεις που έχουμε ήδη ακούσει σε σχέση με τις απειλούμενες γλώσσες. Σίγουρα ε, υπάρχει ένα θέμα ορισμού της απειλούμενης γλώσσας. Ε, θα μπορούσαμε να σπαταλήσουμε πολύ χρόνο για αυτό το θέμα, αλλά εν τέλει μπορεί και να μην ήταν τόσο υποφελές. Αυτά που ακούσαμε για τις νέες τεχνολογίες ε, της ε, ε, πληροφορίας, υπάρχουν δεδομένα, όπως σας είπα και στην παρουσίαση μου, ότι προσφέρει ιδιαίτερα προνόμια, αλλά και αντιπροσωπεύει κινδύνους ταυτόχρονα για τις απειλούμενες γλώσσες ο νέος κόσμος της πληροφορικής. Ε, αυτά τα βλέπουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, ε, όταν γίνονται μελέτες παραδείγματο χάρη στην Αφρική για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, για την προώθηση των μειονεκτικών γλωσσών. Παραδείγματο χάρη με τη δημιουργία νέων λογισμικών που καθιστούν ευχερέστερη τη χρήση αυτών των γλωσσών. Βλέπουμε ότι αυτό είναι υποφελές. Όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε ταυτόχρονα ότι βάσει ε, στατιστικών στοιχείων βλέπουμε ότι μπορεί, μπορούμε να ε, αναμένουμε οικονομικά κέρδη μέσα της χρήσης αυτών των γλωσσών αλλά και της ε, καινοτομία. Η αξία της γλώσσας όμως δεν μετράται μόνο σε χρήματα. Η αξία συνδέεται με παράγοντες όπως η κοινωνική συνοχή και ούτω καθεξής. Θα έπρεπε να συνυπολογίζονται τέτοιοι παράγοντες όταν αποτιμούμε την αξία μια μιας γλώσσας. Σε σχέση τώρα με την θέση της Επιτροπής είναι σημαντικό να ε, στείλετε ηχηρά και θετικά μηνύματα για τη χρήση των μειονεκτικών γλωσσών. Είναι σημαντικός ο ρόλος της δικής σας Επιτροπής ε, σε ρητορικό επίπεδο στην Ευρώπη. Ε, υπάρχει μια ικανή επιχειρηματολογία υπέρ της χρήσης αυτών των μειονεκτικών γλωσσών, όμως αν δείτε στην πράξη τι έχουμε καταφέρει, είναι πενιχρά τα αποτελέσματα. Θα έπρεπε λοιπόν ναι, από τα εύκολα και να περάσουμε στις δράσεις. Ε, αυτά είναι τα λίγο στα σχόλια που κάνω αρχικά μετά από τις παρατηρήσεις που ακούσαμε. Σας ευχαριστούμε. Τώρα, ε, Κλέμεν Φεράντο, αν θέλετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις και εσείς, ε, σύντομα. Πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο καλύτερα αυτό περί οικονομίας και των μη γεμονικών γλωσσών που σας αποκαλούμε. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται εδώ. Έχουμε τη μελέτη ΕΛΑΝ που δείχνουν τη σημασία των μικρότερων γλωσσών στην τοπική οικονομία. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση από ένα μέρος Ευρώπης πάει στη Ρουμανία, στο τμήμα που ομιλούνται τα Ουγγρικά και χρησιμοποιήσει εκτός της Ρουμανικής και την Ουγγρική γλώσσα, τότε θα έχει πολύ περισσότερε δυνατότητε προσέλκυση πελατών από το αν περιοριστεί στα ρουμανικά που είναι η επίσημη γλώσσα του κράτου. Επομένω, ε, ναι, δεν επιτίθεται ε, κατά, η μία γλώσσα κατά της άλλης, ε, αλλά μπορεί να βοηθήσει. Επίσης, μπορούμε να μιλήσουμε για μεθοριακές ή διασυνοριακές γλώσσες. Όπως είπε ο Ισπανός βουλευτής πριν, στην κοιλάδα του Αράν, παραδείγματος χάρη, ή στην Οξυτανία μεταξύ της Κυρίας του Αράν και της Νότιας Γαλλίας της Οξυτάνιας μιλούνται, υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες ε, εκεί. Άρα θα μπορούσαν αυτές οι δύο γλώσσες, αν ε, προσφέρονται ή ε, χρησιμοποιούνται, αυτό να βοηθήσει και να τονώσει την τοπική οικονομία. Ευχαριστώ. κυρία Νίκφορ, τώρα για να δώσω κάποιες σύντομες απαντήσεις, σας ευχαριστώ ακούστηκε η εξή ερώτηση. Τι μπορεί και πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσει η χρηματοδοτική υποστήριξη. Όπω και στο παρελθόν, θα έπρεπε να συνεχίσει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη και τα μέλη ε, προ προσχώρηση να αναλαμβάνουν δράσει υπέρ των μειονεκτικών γλωσσών. Δεν υπάρχει άλλο νομικό εργαλείο ε, προ στιγμή. Είναι μακρά η διαδικασία και μπορεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση τι ε, στη μειονεκτική ψηφική γλώσσα και τη εστί απειλούμενη γλώσσα πρέπει να συνεχιστούν αυτές οι δράσεις. Α, θα ήθελα επίσης να σας παραπέμψω και σε ένα έγγραφο όπου υπάρχει ένας κατάλογος των γλώσσων στον Άτλαντα βλέπουμε τις χώρες μόνο που ε, έχουν επικυρώσει ε, τον χάρτη, δηλαδή για τα καταλανικά βλέπουμε μόνο την Ισπανία, βλέπουμε ε, τις χώρες μέσα σε αυτό το χάρτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση αποκλειστικά και μόνο. Σας ευχαριστούμε κύριος Μόσλη. Τώρα για να κλείσουμε αυτό το γύρο, σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ορισμένα σχόλια τα οποία έγιναν ευθύ εξ αρχή έκαναν τον διαχωρισμό ανάμεσα σε γλώσσε μειονοτήτων και γλώσσες που απειλούνται από εξαφάνιση. Ε, εγώ ε, γνωρίζω πολύ καλά αυτή τη διαφορά που υπάρχει και χαίρομαι που το επισήμαναν και άλλοι σήμερα. Εγώ όταν έκανα προηγουμένω την ομιλία μου, κοιτάξτε, εγώ δεν μίλαγα, δεν αναφέρθηκα ιδιαίτερα στην Ευρώπη, απλά έθεσα το όλο θέμα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ίσως θα έπρεπε να πω ότι ο αριθμός των γλωσσών μειονοτήτων που δεν απειλείται, ο λόγος, ο συσχετισμός με τις άλλες γλώσσες είναι διαφορετικός στην Ευρώπη από τις άλλες υπήρους. Και αυτό θα έλεγα ότι οφείλεται σε διάφορους οργανισμούς και ρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες από διάφορους φορείς οι οποίοι φορείς ε, προσπάθησαν να αναχαιτήσουν τουλάχιστον ε, την διολίστηση γλωσσών που θα μπορούσαν να κατρακυλήσουν σε γλώσσες μειονοτήτων ή γλώσσες απειλούμενες ε, από εξαφάνιση. Υπάρχουν γλώσσες που στην Ευρώπη διατηρούνται πολύ καλύτερα λόγω των μέσων που υπάρχουν και αυτό δεν θα συνέβαινε αν οι γλώσσε αυτέ ομιλούνται σε άλλε υπήρου. Ο εισηγητή λοιπόν τώρα, ο κύριο Αλφόνση. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ποιο ε, βαθμό μπορώ να σας εξηγήσω ε, ήδη από τώρα πώς θα ε, ποιο πρίσμα είναι το, ε, το, πυρήνα και η προσέγγιση τη εκθέσης μου. Ξεκινώ από τη διαπίστωση, την πεποίθηση ότι όλες οι γλώσσε αποτελούν κληρονομιά της Ευρώπης. Η πολυμορφία άλλωστε είναι σλόγγαν στην Ευρώπη και πιστεύω ότι πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία και με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους. Μεταξύ αυτή λοιπόν και η διάσταση της γλωσσική και πολιτιστική ή πολιτισμική πολυμορφία. όταν οι ιδρυτές ε, πατέρες ε, τη δεκαετία του 50 έθεσαν τα θεμέλια. Έγινε αντιληπτό ότι είναι πλούτος η πολυμορφία της Ευρώπης. Τώρα, έχουμε αυτέ τι μειονοτικέ γλώσσε, όπω τα ογκρικά στη Ρουμανία. Από ευρωπαϊκή πλευρά δεν κινδυνεύει αυτή η γλώσσα σίγουρα, γιατί η πρακτική και η άσκηση της, ε, του πολιτισμικών δραστηριοτήτων διατηρούν αυτή τη γλώσσα στη Ρουμανία. Τι θέλουμε όμως να προωθήσουμε για τον Ευρωπαίο πολίτη. Ουσιαστικά θέλουμε να προωθήσουμε τη γλωσσική πολυμορφία, ώστε άνθρωποι που λόγω της ιστορίας τους ε, στη χώρα τους έχουν φυσική πρόσβαση στη μητρική τους γλώσσα ε, και εμπλουτίζουν τελικά την γλωσσική κληρονομιά. Ο παππούς μου ήξερε κορσικανικά και γαλλικά, ε, ήταν γονός ενός αγρότη, αναλφάβητου. Και έλεγε ότι τελικά οι Κορσικανοί ε, μάθαιναν πολύ πιο καλά και τα γαλλικά και μπορούσαν να έρθουν σε επαφή και με τους Μαροκινούς. Δηλαδή έχουν μια φυσική ευχέρεια ε, και ευκολία. Την επιβεβαιώνουν και οι επιστήμονες. Η δίγλωση, αυτή που είναι φυσικά δίγλωση λόγω της ε, οικογενειακής τους ιστορίας. Αυτή μπορούν να είναι πολύγλωση στο μέλλον και στις επουδές τους και αργότερα στον επαγγελματικό τους βίο. Αυτό λοιπόν συνιστά δυνητικά ένα έναν γλωσσικό πλούτο. Αυτό θα εφαρμοστεί και στις μειονοτικές γλώσσες που μιλούνται βέβαια σε ανταγωνισμό με μια άλλη γλώσσα. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε το στόχο της γλωσσικής πολυμορφίας. Αυτό το βλέπουμε από την πλέον νεαρή ηλικία, από την τρυφερή ηλικία του παιδιού. Και είναι σημαντικό να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και θα μπορούσε βέβαια και το πρόγραμμα που έχουμε ήδη να ε, επεκταθεί, αλλά πιστεύω ότι και το έρασμος που βοηθάει δηλαδή Έλληνες φοιτητές στη Γερμανία, όλα αυτά συνεισφέρουν ε, στην ε, πολυγλωσία και των Γερμανών, να μάθουν ελληνικά για παράδειγμα, αν αυτό βέβαια ενδιαφέρει και τους γονείς και η ιδέα ότι η πολυγλωσία, μάλλον η γλωσσική πολυμορφία, η φυσική γλωσσική πολυμορφία που αποκτάται από τη γέννηση είναι ένα θεμελιώδε στοιχείο για την γλωσσική πολυμορφία, νομίζω ότι αυτή δεν είναι σημαντική και όλου μα πρέπει να μα ενδιαφέρει. Έχουμε λοιπόν έναν, ένα κίνητρο, έχουμε αυτή την πτυχή ότι αποτελούν κληρονομιά όλε οι γλώσσε και έχουμε και μέτρα να υιοθετήσουμε που πιστεύω θα πρέπει να υπερβούν και υπερβαίνουν ουσιαστικά τις ε, γλώσσε που απειλούνται με εξαφάνιση. Έχει να κάνει και με τι μοτικέ γλώσσε και με την ίδια την πολυμορφία και με τις επίσημες γλώσσες. Ο προς το συμφέρον όλων αυτών των γλωσσών είναι. Ε, ακόμα και αυτών που είναι κυρίαρχες, επικρατούν δηλαδή λόγω ε, και τη κατάσταση και κάποια θεσμική ενδεχομένω προτίμηση. Σίγουρα είναι εξελικτική η κατάσταση και στι γλώσσε και στα κράτη και σήμερα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση διαφορετική από αυτή ε, τη δεκαετία του 80 όταν συζητήθηκε ακόμη και στην Επιτροπή μα εδώ ο χάρτη των γλωσσών. Είναι σαφές ότι οι κίνδυνοι που απειλούν σήμερα γλώσσε μπορούν να διαφέρουν. Στο παρελθόν ήταν η πολιτική καταστολή που απειλούσε τις γλώσσες, ε, είναι προφανές. Σήμερα φυσικά και αυτό δυστυχώ μπορεί να υφίσταται ακόμη και στην Ευρώπη, ε, πρέπει λοιπόν η πολιτική καταστολή να φροντίσουμε να πάψει. Αλλά αύριο η ψηφιακή πρόοδο τη τεχνολογία, όπω είπε και ο συνάδελφο, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τι γλώσσε. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι και οι κίνδυνοι είναι εξελικτικοί, μεταλλάσσονται και επίσης και οι ε, καταστάσεις αλλάζουν. Και ο Φύσης μίλησα για τα βασικά, που είναι μια από τις σπάνιες γλώσσες για τις οποίες μπορούμε να πούμε ότι από το 80 και μετά είναι καλύτερη η κατάστασή της σε σχέση με το παρελθόν. Μπράβο στους Βάσκους που τα κατάφεραν. Αλλά για μια γλώσσα που είχε μια θετική εξέλιξη έχουμε 10, 20, 30 ή 80 που δυστυχώς υποβαθμίστηκαν έτσι περαιτέρω, που είναι αρνητικές, ε, η αρνητική εξέλιξή τους. Έχουμε λοιπόν αυτή την προσέγγιση, κληρονομιά, άρα ε, πλησιάζουμε και στην επιστημονική προσέγγιση και στην προσέγγιση της UNESCO. Πρέπει να ε, έχουμε τα κατάλληλα κριτήρια, θα θεσπιστούν αυτά τα κριτήρια και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει στην ανάπτυξη του εργαλείου αυτού και τη διατήρησή του. Για μας όμως που είμαστε μια πολιτική, ένα πολιτικό θεσμό, πρέπει να έχουμε πολιτική προσέγγιση. Μια γλώσσα λαμβάνεται υπόψη από τη στιγμή που η γλωσσική κοινότητα κάνει το σχετικό αίτημα, προτείνει ένα σχέδιο δράση, προτείνει ορισμένα μέτρα και ζητά βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το έργο αυτό που δεν είναι μόνο για την ίδια την γλωσσική αυτή κοινότητα, αλλά και για όλη την ευρωπαϊκή κληρονομιά, όπως είπα. Για τις δράσεις τώρα, στην έκθεσή μου θα προσπαθήσω να μπω σε λεπτομέρειες και να κάνω και κάποιες προτάσεις. Αλλά από ό,τι ακούσαμε στις παρεμβάσεις των εμπειρογνωμόνων μας, αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι ναι, μέχρι το 2000 είχαμε ένα προπολογισμό, είχαμε κάποιες δράσεις, άρα ε, δραστηριοποιούμασταν ως Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις απειλούμενες γλώσσες. Από το 2000 και μετά έπαψε να υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Και στην έκθεσή μου ελπίζω να δώσω κίνητρα ε, για να επανενεργοποιηθεί μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των γλωσσών και της υποστήριξης της απειλούμενης κληρονομιάς. Θα ήθελα λοιπόν ε, να μάθω κατά πόσον ε, ο κύριος Τομάζη, εκπρόσωπος Κομισιόν, είναι παρόν ή όχι. Παρακαλώ κύριε Τομάζη, έχετε το λόγο. Θέλω να σας πω ότι εγώ παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες αυτές τις ε, παρεμβάσεις και κατανοώ βέβαια αυτά που είπε ο κύριος Αλφόνση και κατανοώ πολύ καλά το ότι είναι δύσκολο για την Επιτροπή να βρει μια νομική βάση για να στηρίξει τις ε, γλώσσες ε, που απειλούνται με αφανισμό, κυρίως όσον αφορά τις γλώσσες ε, που δεν είναι επίσημες στα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή λοιπόν καταλήγει στην λύση των δικτύων για να στηρίξει αυτές τις γλώσσες δίκτυα λοιπόν για να προάγουν την ε, γλωσσική ποικιλομορφία. Ακούσαμε σήμερα ένα παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, δίκτυα για τις γλώσσες που αντιμετωπίζουν, που βρίσκονται σε πρόβλημα και αντιμετωπίζουν κινδύνους. Η Επιτροπή οργανώνει επίσης μία πλατφόρμα για την κοινωνία των πολιτών, για την πολυγλωσσία και εκεί προβλέπονται μία σειρά συστάσεων που αφορούν ε, όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη χωρίς καμία διαφοροποίηση. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα προγράμματα. Δεν υπάρχει μόνο το πρόγραμμα της ε, διαβίου μάθησης, αλλά υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες ε, που στηρίζουν τις περιφερειακές γλώσσες, παραδείγματο χάρη πρωτοβουλίες για την λογοτεχνική μετάφραση από αυτές τις γλώσσες και προς αυτές τις γλώσσες. Κατά τα άλλα, συνεργαζόμαστε και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και σε αυτόν λοιπόν τον τομέα προσπαθούμε να προάγουμε την ε, γλωσσική ε, ποικιλομορφία. Σήμερα, βεβαίως αυτή η έννοια έχει διαφορετική, διαφορετικό νόημα. Και θέλω να σας πω ότι με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να δω ε, το τι θα περιλαμβάνει αυτή η έκθεση προς την Επιτροπή και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς θα τα λάβουμε όλα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και κάτι ως γλωσσολόγος. Πολύ σημαντικό αυτό που υποστήριξαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, ότι δηλαδή οι γλώσσες που αντιμετωπίζουν κινδύνους, αυτοί είναι ζώντες οργανισμοί. Δεν είναι... Ε, Αποκρισταλωμένε οντότητες που μπορεί κανείς ε, να τις διατηρήσει σε ένα μουσείο. Και εφόσον μιλάμε για ζωντανές οντότητες, αυτές εξελίσσονται, διότι οι επαφές είναι όλο και πιο στενές. Άρα δηλαδή υπάρχει μια δυναμική που πρέπει να την ερευνήσουμε και να έχουμε κατά νου ότι οι γλώσσες αυτές είτε είναι μικρές είτε μεγάλες, είτε αντιμετωπίζουν κίνδυνο ή όχι, οι γλώσσες αυτές ε, θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Και αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε μια μια φυσιολογική και όχι τραυματική εμπειρία όπως ε, θα μπορούσε να είναι η εξαφάνιση μιας γλώσσας και αυτό το γεγονός ε, θα αποδυνάμωμε, θα καθιστούσε πιο φτωχιά την ε, δική μας την πολιτιστική κληρονομιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την Επιτροπή και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Αλφονσί θα παρουσιάσει την έκθεσή του τον Απρίλιο και θα ψηφιστεί τον Μάιο. Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα της μυρίσιας διάταξης, στο σημείο υπαριθμών 5. Εκεί προβλέπεται η ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του Δικτύου Εκδοτών Εφημερίδων Press Europe. Είναι ένας οργανισμός με έδρα το ε, Παρίσι και κάθε μέρα ε, παρουσιάζει ένα απάβγασμα ε, από διάφορες δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, μεταφράζεται σε πάρα πολλές γλώσσες αυτό το απάβγασμα ε, και ιδρύθηκε το 2009 ε, με τη συνεργασία τεσσάρων εξειδικευμένων εφημερίδων περιοδικών του Παρισιού, Κοριέρε του Παρισιού, της Λισαβόνας, της Βαρσαβίας και την τη της Ρώμης. Ε, βέβαια, το δίκτυο αυτό ε, στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά, έχει διατηρήσει την ε, συντακτική της ανεξαρτησία και έχει και σχετικό ιστότοπο στο διαδίκτυο. Μέχρι τις 11.45 ε, έχουμε χρόνο για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τους ομιλητές να λάβουν το λόγο, αλλά ή δυνατόν να μην υπερβεί κανένας από αυτούς τα 10 λεπτά και να μας παρουσιάσουν σύντομα τις εργασίες αυτού του φορέα. Και κατόπιν θα δώσω το λόγο σε εσά για ερωταπαντήσεις. Ε, η πρώτη παρέμβαση ε, είναι του κυρίου Πολ Σέιν. Καλημέρα. Κύριε Αντιπρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα ε, να συστηθώ. Είμαι συντονιστής ε, στο Press Europe ε, από το 2009 και μετά. Επίσης για πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο στόχος είναι με αμεροληψία, με ανεξαρτησία να αναμεταδίδονται στη διεθνή ιδιοσιογραφία ε, τα όσα διαμείβονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορες γλώσσες όπως γαλλοαγγλικά, ε, γερμανικά, πολωνικά, ρουμανικά, πορτογαλικά και ούτω καθεξής. Ε, το περιεχόμενο διαθέσιμο σε όλες αυτές τις γλώσσες 10 είναι στον αριθμό συνολικά και το ίδιο ισχύει και για τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε το συντάκτη μας εδώ, την εκπρόσωπη πρόσωπο του Ιντερνασιονάλ από τη Ρώμη, ε, επίσης το συντονιστή του γερμανικού τύπου, ε, την κυρία Γιουντίτ Σινίτσε που ε, είναι επικεφαλής της Ολλανδικής εκδοχής της του ιστοτόπου μας. Η πρόεδρος μας προσκάλεσε εδώ και την ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον Αντιπρόεδρο για την παρουσίαση που έκανε και την πρόσκληση που μας απίθυνε για να σας παρουσιάσουμε το Press Europe. Ποιο είναι ο στόχο αυτού του σχεδίου, Βασιστήκαμε στην εξή ε, διαπίστωση. Ο δημόσιο διάλογο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά υπάγεται σε εθνικά πρότυπα και αυτό αντιβαίνει ε, στο πνεύμα τη Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Όταν μιλάμε για την Ευρώπη, συχνά βλέπουμε από την εθνική μα οπτική γωνία τι προκλήσει τη Ευρώπη. Όμω, η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια οικογένεια γεννάται από την αντιπαράθεση των ιδεών σε ένα κοινό χώρο, ούτω ώστε να αντιληφθούμε ποιο είναι το νόημα μιας άποψη που είναι διαφορετική από τη δική μας. Πρόκειται για ανταλλαγή ιδεών λοιπόν στον ευρωπαϊκό χώρο. Πώς να κατανοήσουμε ε, όμως ε, τους υπολείπους Ευρωπαίους όταν δεν ε, μιλούμε τη γλώσσα τους. Πώς να κατανοήσουμε τους πολίτες μιας άλλης χώρας αν δεν ζω και εγώ δεν έχω τα ίδια βιώματα καθημερινά. Χάρη στο διαδίκτυο, αυτός είναι ο στόχος του Press Europe, να πλησιάσουν οι Ευρωπαίοι, να ανταλλάξουν μαρτυρίες και βιώματα και να πλησιάσουν ένα τον όλον. είμαστε μοναδικοί στο είδος μας, διότι δωρεάν προσφέρουμε στους αναγνώστες μας σε μια πλουραλιστική ειδησεογραφία, ιδιαίτερα ποικιλόμορφη, χάρη στην οποία οι αντιπαραθέσεις ε, ε, ε ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες εξαλείφονται και γινόμαστε Ευρωπαίοι. Πάνω από 2.000 άρθρα δημοσιεύονται σε 10 ε, γλώσσες. Πάνω από 1.500 δημοσιογράφοι, ερευνητές, συντάκτες, δημοσιεύουν άρθρα στην ιστοσελίδα μας. 10.000 επισκέψεις έχει ο ιστότοπός μας, έχει αυξηθεί ε, πάρα πολύ ο αριθμός των επισκεπτών ε, στα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επίσης ε, και στην εκδοχή του ιστοτόπου για τα κινήτα. Για κάθε ένα από τα άρθρα έχουμε πάνω από 40 σχόλια. Ε, η συσπήρωση των Ευρωπαίων μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, μέσα από πολύγλωσσα σχόλια, από δημοσκοπήσεις ε, που δημοσιεύουμε στην ε, ιστοσελίδα, με πολύ αυτό τρόπο προσεγγίζουν ο ένας τον άλλον οι Ευρωπαίοι. Οι διανοούμενοι, οι πολίτες, οι ακαδημαϊκοί, όλοι όσοι θέλουν να μιλήσουν για την Ευρώπη και να ανταλλάξουν τις ιδέες τους, συγκεντρώνονται και συνευρίσκονται στον ιστότοπό μας. Ε, ε, είμαστε στο, ε, στην καρδιά ενός πολύγλωσσου δικτύου, είμαστε χώρο συναισθίασης αυτών που θέλουν να ακουστεί η φωνή τους στην γυραιά Ήπειρο. Έχουμε μια κοινότητα αναγνωστών που συζητούν και σχολιάζουν αυτά που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές τη Ένωση φυσικά, αλλά και τα γεωπολιτικά παγκόσμια διακυβεύματα, τις δημογραφικές εξελίξεις, τις κοινωνικές, κοινωνιολογικές εξελίξεις, αλλά και σχόλια για την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας από το Δουβλίνο μέχρι την Αθήνα. Σας ε, καλώ να διαβάσετε τα σχόλια, να μετάσχετε και εσείς ήδη στη γλώσσα σας, ε, ε, να γράψετε σχόλια στην, στον ιστότοπό μας, ώστε να διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Οι, οι μελλοντικέ ευρωπαϊκές εκλογές το Μάιο του 2014 είναι μια μοναδική ευκαιρία σε παγκόσμια κλίμακα και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Όμως γεννώνται και ερωτηματικά θα συζητήσουμε με πολλούς βουλευτές, με πολλούς δημοσιογράφους, όλοι φοβούνται όμως την αποχή. Υπάρχει αυτός ο κοινό φόβος λόγω της οικονομικής κρίσης, της παγκοσμιοποίησης, της αναδίπλωσης στην εθνική ταυτότητα, η υπεράσπιση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολλά θέματα μας απασχολούν, αλλά δεν είναι ο στόχος της σημερινής παρουσίας. Θέλω μόνο να σας πω ότι υπάρχει ανοιχτή Ευρώπη, δημιουργική Ευρώπη που θέλει να μετάσχει σε αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο την προπόθεση ότι θα έχει τα απαιτούμενα μέσα. Λοιπόν, το διαδίκτυο είναι το πρώτο ε, για την ηλικία 18 ως 35 και η, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ε, δημοκρατικό μέσο ε, με τρόπο ώστε να είμαστε κοντά στους Ευρωπαίους και κυρίως στους νέους Ευρωπαίους που είναι οι μελλοντικοί Ευρωπαίοι. Εν κατακλείδη, η Press Europe ε, θα τραβήξει το ενδιαφέρον των αναγνωστών της εν των εκλογών εκλογών του 2014. Ε, στον ιστότοπό μας θα προωθήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ευρωπαϊκές εκλογές ε, με κυρίους αποδέκτες ε, τους νέους και όσους έχουν μετάσχει στο σχέδιο Εράσμους. Θα ε, βοηθήστε μας και εσείς ε, μέσω των δικών σας δικτύων να προωθήσουμε το Press Europe. Όλοι μιλάνε για δημοκρατική κρίση. Εμείς όμως ε, το διαψεύδουμε καθημερινά ήδη από τώρα πόσο πλούσια και ζωντανή είναι η συζήτηση και πολύγλωση είναι η δημόσια συζήτηση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον συνάδελφό. Madame la Présidente. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, κυρίες και κύριοι Αντιπρόεδροι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Λέγομαι Ενρίκ Μωρίς και είμαι αρχισυντάκτης ε, του Press Europe, 12 ε, δημοσιογράφους, 2 webmaster, 15 ταποκριτές και περίπου 60 μεταφραστές όλη την Ευρώπη απαρτίζουν το προσωπικό μας. Πριν σας παρουσιάσω την λειτουργία του Press Europe, όπως είπε και ο προλαλής σας συνάδελφος, πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά το site μας ε, ε, αποτελεί μία εικόνα του πώς αντιλαμβανόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελείται από 27 χώρες. Άρα πρέπει να παρουσιάσουμε την επικαιρότητα σε όλες τις ε, χώρες. Ποια είναι η συντακτική μας γραμμή. Προτείνουμε με αμερόληπτο τρόπο, με πρωτότυπο τρόπο, ε, πληροφορίες, ε, απόψεις, ε, ενδιαφέροντα, ρεπορτάζ, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες, τόσο στη δική μας Ήπειρος, ο και αλλού. Διαλέγουμε τι διαβάζουν οι πολίτες, μεταφράζουμε τα άρθρα σε 10 χώρες για να μπορούν να τα διαβάζουν και οι πολίτες άλλων χώρων στις δικές τους γλώσσες. Η Press Europe είναι το μόνο μέσο, για παράδειγμα, που οι Γερμανοί μπορούν να διαβάζουν αυτό που διαβάζουν οι Έλληνες. Που μπορούμε να μάθουμε τι διαβάζει κανείς στην Ουγγαρία για τον Μπέμπε Γκρίλο, παραδείγματο χάρη, ή τι θα επιπτώσει θα έχει ένταξη κορατία ε, στην Ένωση ή οικονομικέ συζητήσει που γίνονται χώρα σε διάφορε χώρε. Όλα αυτά τα θέματα μα ε, τα καλύπτουμε. Προτείνουμε διαφορετικέ απόψει για να μπορέσει και ο πολίτη να διαμορφώσει τη δική του άποψη. Εδώ και τέσσερα χρόνια η ομάδα μα επιλέγει, μεταφράζει άρθρα από 400 εφημερίδε περίπου. Προτείνουμε άρθρα από όλη την Ευρώπη, Άρα ουσιαστικά ε, δημιουργούμε προβληματισμό ε, και πιστεύουμε ότι έτσι ανθεί και η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Για παράδειγμα, όταν η Press ε, Europe προτείνει για τους αναγνώστες της Νότιας Ευρώπης άρθρα από την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις σκανδιναβικές χώρες και όταν οι αναγνώστες όλων αυτών των περιοχών ανταλλάσσουν ουσιαστικά απόψεις και εμπειρίες στο μισθό τοπό μας, βλέπουμε να αναδύεται έτσι μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Κάθε άρθρο 50 φορές περίπου σχολιάζεται. Χάρη στο σύστημα αυτόματης μετάφρασης των σχολείων το οποίο αναπτύξαμε στο Press Euro μπορούν οι αναγνώστες μας να καταλάβουν ένα τον άλλο και να ανταλλάξουν απόψη χωρίς το φράγμα της γλώσσας που πολύ συχνά ε, χωρίζει στους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, άρα δημιουργείται μια κοινότητα Ευρωπαίων πολιτών στο site μας. Αυτό το οποίο διαπιστώνω και θα ήθελα να σας μεταφέρω σε εσά τους ε, εκλεγμένους προσώπους των ε, Ευρωπαίων πολιτών ότι υπάρχει μεγάλη τάση για συζήτηση των ευρωπαϊκών θεμάτων και των εθνικών. Όταν αναλύουμε συζητήσεις ε, στο, στον τόπο μας βλέπουμε ότι υπάρχει μια περιέργεια την Ευρώπη η οποία εξηγείται κυρίως γιατί οι άνθρωποι θέλουν να, έχουν μια άλλη επίδραση με το υπερεθνικό αυτό επίπεδο. Και Υπάρχει ένα μεγάλο αίτημα δημοκρατίας, το οποίο διέρχεται μέσω της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ από τη μια του Ευρωκοινοβουλίου και από την άλλη των εθνικών κρατών μέλων και των συμφερόντων που υπηρετούν. Αυτή η ευρωπαϊκή ταυτότητα μπορεί να ενισχυθεί αν οι κάτοικοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στη διάθεσή του μέσα που θα του επιτρέπουν να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Από το 19ο αιώνα η ελευθερία έκφραση στο δικαίωμα στην ενημέρωση εγγυώνται τι αξίε πάνω στι οποίε εδράζεται η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το δικαίωμα ψήφου είναι επίση πυλώνα αυτή τη ταυτότητα με τη δημοσίευση απόψεων, γνωμών, με ευαισθησίε εφορτικών χωρών. εξασφαλίζουμε τη διασύνδεση αυτών των δύο δημοκρατικών απαιτήσεων Έρχομαι τώρα ε, στο διαδικτυακό μέσο, το διαδικτυακό μέσο, που φυσικά δεν είναι η πανάκια για την προσέγγιση των ευρωπαϊκών πολιτών, αλλά είναι το πρώτο ε, μέσο Ενημέρωση μεταξύ των νέων. Το είδαμε με την προεκλογική στρατεία του Μπαράκ Ομπάμα στη ΣΥΠΑ, αλλά και πρόσφατα στην Ιταλία με την επιτυχία του Μπέπε Γκρίλο και βλέπουμε πόσο μοναδικό είναι το ίντερνετ και γι' αυτό το Press Europe ε, εκτός της ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο έχει και κάποιες ε, κινητές εφαρμογές ε, και επίσης τα δίκτυα τα κοινωνικά, το Google, το LinkedIn, το Twitter και όλα αυτά επίση επενδύει το Press Europe που είναι ένα ψηφιακό μέσο αναφοράς για την ε, επικαιρότητα είναι και ένας τόπος μετάλλαξης. Ε, αλλάζουμε κι εμείς για να μπορεί να επικοινωνεί καλύτερα ο ένας Ευρωπαίος πολίτης με τον άλλο. Και θα δώσουμε μεγάλη προσοχή ε, σύντομα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εκλογές. Το 2009 όταν έγιναν οι τελευταίες ευρωεκλογές εμείς δεν είχαμε τα ίδια εργαλεία που έχουμε σήμερα, άρα μπορούμε να βασιστούμε στα τέσσερα χρόνια ε, εμπειρίας και ξέρουμε όπως και εσείς ότι στις εκλογές δύσκολο να κινητοποιηθεί πολλοί κόσμος και να πάει να ψηφίσει στις κάλπες. Εμείς θέλουμε όμως να πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ότι θα πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Πέραν αυτής όμως της προθεσμίας του 2014 Έχουμε και το μοντέλο πολιτικής συμμετοχής το οποίο εξελίσσεται, άρα πρέπει να ανακαλύπτουμε, να εφεύρουμε νέες μορφές ε, ε, διαρκούς επικοινωνίας ε, των βουλευτών και των ψηφοφόρων τους. Θα καλέσουμε λοιπόν ευρωβουλευτές στις εκδηλώσεις μας και όλες αυτές οι εκδηλώσεις θα μεταδίδονται στο ίντερνετ απευθείας. Θα υπάρχει λοιπόν δυνατότητα αλληλεπίδρασης, διάδρασης. Αυτό θα το κάνουμε από φέτος, το 2013 και μέχρι τις ευρωεκλογές του 2014. Θα καλέσουμε επίσης και τους αναγνώστες και τους σχολιαστές, τους πιο ενεργούς, για να σας ε, να επικοινωνήσουν απευθείας με εσά. Πρώτη συζήτηση, σας το λέω ήδη, 4 Ιουνίου, την Τρίτη, εδώ στο Κοινοβούλιο, στο Voxbox. Θα υπάρχουν εκεί ευρωβουλευτές, προσωπικό Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκέπτες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα σταυροδρόμι αυτός ο χώρος εκεί. Τέλος, θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα απαραίτητο θεσμικό όργανο για τη ε, δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ε, διαλόγου ε, που θα είναι κατά την, και, κατά την παράσταση και δημιουργικός. Θέλουμε να είμαστε σύνδεσμος μεταξύ των διαφορετικών απόψεων. Θέλουμε στους αναγνώστες μας να προσφέρουμε μια καλύτερη κατανόηση για την Ευρώπη και το μέλλον της. Άρα εκφράζω σε εσά την ευχή σήμερα να μπορέσουμε να ε, παρακολουθήσουμε και να εμψυχώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις συζητήσεις και τις εργασίες σας μέχρι τις εκλογές του 2014. Σας ευχαριστώ πολύ και θα δώσω τώρα το λόγο στον Αλισάντρο Παβέντα, τον πρόεδρο του Ιντερνατσιονάλ. E Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Τώρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα να τεθούν ερωτήσεις. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη ε, και γι' αυτό σας κάλεσα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουν λεχθεί. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα κατά νου και το χρόνο. Συνάδελφοι, ποιος λοιπόν επιθυμεί να λάβει το λόγο? Ο Μόρτον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη δουλειά που κάνατε. Βεβαίως, εγώ είχα την ευκαιρία να σας συναντήσω προηγουμένως και να μιλήσουμε για τις ε, προσπάθειες που κάνετε και νομίζω ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ είμαι ένας από τους ε, οπαδούς σας. Ε, νομίζω έχετε και πάρα πολλούς άλλους βέβαια και έχω μπροστά μου τον υπολογιστή μου και τη δυνατότητα να σας παρακολουθώ και να το κάνουν και άλλοι τους, το συστήνω. Γιατί πραγματικά εδώ πρόκειται για έναν από τους ε, τομείς ε, όπου μπορούμε ε, να επιτύχουμε έναν πραγματικό ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο. Σας συγχαίρω λοιπόν. Σαφώς και ζείτε επικίνδυνη ζωή με την έννοια ότι στηρίζεστε οικονομικά από όλους αυτούς τους θεσμούς και έχουμε κάποιες ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε και επειδή είσαστε εδώ θα ήθελα να μου επιτρέψει να σα κάνω κάποιε ερωτήσει. Αυτός ο χάρτη ε, που έχετε παρουσιάσει ε, είναι πολύ παραστατικός και ενημερωτικός ε, αλλά φοβάμαι ότι εδώ ξεχάσατε τις σκανδιναβικές χώρες τα σκανδιναβικά μάλλον έχετε ακόμα και τα ρουμάνικα και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής. Θα ήταν ε, πολύ σημαντικό να ε, κατακτήσετε και τις σκανδιναβικές χώρες. Νομίζω ε, πολλοί πολίτες στη Σκανδιναβία θα ενδιαφερόντουσαν ιδιαίτερα να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις που γίνονται στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Απλά έτσι αυτό είναι μια φιλική συμβουλή. Και ένα άλλο θέμα. μεταφράζεται και ε, αναπαράγεται άρθρα σε εφημερίδες. Αλλά τι γίνεται με τις εικόνες. Τώρα πλέον υπάρχει εξή κατάσταση. Κατά τα επόμενα χρόνια ε, πάνω από 90% των πληροφοριών θα είναι εικόνες. Και είπατε ότι είναι φιλοδοξία σας ε, να έχετε απήχηση στους νέους. Επειδή λοιπόν οι νέοι σήμερα αποκτούν σχεδόν όλες τους τις πληροφορίες ε, από ε, εικόνες, από το διαδίκτυο και την τηλεόραση, μήπως ε, έχετε έτσι κάποια ιδέα του πώς μπορεί κανείς να διεισδύσει σε αυτό το χώρο. Και τέλος, επιτρέψτε μου μια ερώτηση που αφορά στις εκλογές του επόμενου έτους. Έχετε κάποια συγκεκριμένη ιδέα για το πώς προτίθεστε να ε, καλύψετε του χρόνου τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Ταβάρης. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πορτογαλική καμπίνα σήμερα. Είμαι αναπληρωτής εδώ και δεν προσφέρεται αυτόματα η μετάφραση. Θα μιλήσω γαλλικά σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όσα έχετε κάνει. Είμαι τακτικός αναγνώστης του Press Europe και ξέρω ότι η πορτογαλική εκδοχή ε, χρησιμοποιείται και εκτός Πορτογαλίας. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον για όλους όσους ε, παρακολουθούν την ευρωπαϊκή επικαιρότητα στη Βραζιλία, στην Αφρική με την κρίση. Έχουμε όλα ένα και περισσότερους Πορτογάλους παραδείγματο χάρη το ίδιο. Ισχύει και για την αγγλική εκδοχή και τη χρήση της στη ΣΥΠΑ παραδείγματο χάρη σε blog, σε ιστολόγια οικονομικού χαρακτήρα κυρίως το έχω δει σχετικά στοιχεία. Σα Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τις ε, εκλογές, ε, τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 θα ήθελα να σας θυμίσω ότι εγκρίναμε πέρυσι ένα ψήφισμα για τις εκλογές Και ήθελα λοιπόν ε, να πω ότι κάποιες ε, τροπολογίες δεν είναι ξεκάθαρες ε, και χωρίς τη βοήθειά σας θα δυσκολευτούμε να προωθήσουμε τις ιδέες μας. Ποιοι θα είναι υποψήφοι σε επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Θέμα χέρια σημασίας για ένα δημοκρατικό ε, καθεστώς και δεν μιλώ μόνο για τους αιρέτου, μιλώ και για την εκτελεστική εξουσία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό θα ήταν σημαντικό να συμβαίνει σε μια, ένα δημοκρατικό χώρο. Ε, σε σχέση με τις προγραμματικές δηλώσεις, οι υποψήφοι, οι επίτροποι, αν έχουν πρόγραμμα, γιατί δεν είναι και δεδομένο, μπορεί να βασίζονται μόνο στην ισχύ των συνασπισμών τους ε, που έχουν είτε στο Κοινοβούλιο είτε στο Συμβούλιο, Προτείναμε λοιπόν ε, αυτή την ιδέα, δεν προβλέπεται φυσικά στην νομοθεσία, είναι μια σύσταση. Ζητούμε προγραμματικέ δηλώσει από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πέραν αυτού, και αυτό είναι πολύ καλό, διότι έχουν μεταφραστεί αυτέ οι ιδέε για να, γίνονται, ε, για να γίνεται ένα δημόσιο διάλογο ανάμεσα στου υποψηφίου, να υπάρξει αντιπαράθεση δηλαδή των ιδεών του. Και αυτό είναι σημαντικό. Άλλο εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι να κάνουμε μια πραγματική Ευρωπαϊκή Προεκλογική Εκστρατεία. Έχουμε καταθέσει μια τροπολογία βάσει της οποίας ε, καλούνται υποψήφοι επίτροποι προσωπικά να παρουσιάσουν ε, το πρόγραμμά τους ε, στις 27 και μελλοντικά 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό γιατί πολύ ε, ευκολότερο είναι να κάνει κάποιο σε μια ευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία αρχίζοντας από την Αθήνα παραδείγματος χάρη. Ε, ένας υποψήφιος επίτροπος ε, πρέπει να πάει στην Αθήνα να εξηγήσει στους Έλληνες με ποιο τρόπο πιστεύει ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε το ευρωπαϊκό αρχικά πρόβλημα και στη συνέχεια το ελληνικό. Για να γίνει αυτό, Χρειάζεται ένα ε, καλό δίκτυο δημοσιογράφων, ε, ιστοτόπων, ε, τηλεοπτικών δικτύων, ε, ραδιοφωνικών σταθμών, όπου θα διεξάγεται αυτός ο δημόσιος διάλογος πριν από τις εκλογές, με τρόπο ώστε να προετοιμάσουμε και το δημόσιο διάλογο στις πρωτεύουσες, στις φοιτητικές αιστείες, στα πανεπιστήμια, παντού. Ε, πρέπει να είμαστε ευρηματικοί. Ε, οι υποψήφοι ε, στις αμερικανικές εκλογές πριν από έναν αιώνα μέσα στα τρένα κάναν την προεκλογική τους εκστρατεία. Πολύ οικολογικός τρόπος για να κάνει κάποιος προεκλογική εκστρατεία. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να είμαστε ευρηματικοί με τρόπο ώστε να ακουστεί η φωνή των υποψηφίων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό θα τονώσει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή δημοκρατία, το ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο. Ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν μπορούμε όμως τώρα να χρησιμοποιήσουμε την Press Europe ε, ως όχημα δικό μας ε, για την ε, προεκλογική εκστρατεία. Βεβαίως και μπορείτε να ενημερώνετε και προφανώς μπορείτε να κάνετε προεκλογική εκστρατεία για όλους. Μπορείτε να κάνετε και για μένα. Αλλά μην ενισχύετε, εγώ δεν θα ξανά είμαι υποψήφια. Τέλος. Χαίρομαι που σας γνώρισα και διαβάζω αυτά που γράφετε για την Αφρική, ιδιαίτερα θετικά και πολύ καλό αυτό που έκανε η Κομισιόν. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση δεν συμβαίνει πάντα αυτό, αλλά σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει μια επιτροπή η οποία παρουσιάζει διάφορα θέματα και κάτω από διαφορετικό πρίσμα. Ε, Παραδείγματο χάρη, βλέποντα αυτά που λέτε τώρα για την Κύπρο, που ε, παρουσιάζεται το πώ ε, το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Κύπρο. Αυτό νομίζω ότι πραγματικά δίνει μια εικόνα τις ε, πολυμορφίες που υπάρχει και ε, ανάλογο και κάτω από ποιο πρίσμα το βλέπει ο καθένας. Ε, χαίρομαι που μιλήσαμε σήμερα μαζί σας ε, στο πλαίσιο των απειλούμενων με εξαφάνιση γλωσσών. Ε, βεβαίως και δεν θεωρώ ότι θα έχετε αναφορές και άρθρα σε κορσικά, στα αλσατικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Ίσως όμως θα μπορούσατε, όπως είπε και ο να καλύψετε αυτή την λευκή κοιλίδα που υπάρχει στο χάρτη. Έχω την εντύπωση ότι οι σκανδιναβικές χώρες πολλές φορές είναι πιο ψύχρεμοι, πιο νυφάλιοι, ε, τουλάχιστον όχι τόσο παρορμητική όσο οι νότιοι. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, όπως είπε και ο άλλο, έχετε τη Ρουμανία, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχετε την Ουγγαρία. Και σήμερα η Ουγγαρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι μεταξύ άλλων το πρόβλημα των Ούγγρων είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα τους και πολλά από αυτά που κάνουν οι Ούγγροι. Γι' αυτό το λόγο ε, σε εμά δεν γίνονται κατανοητά, γιατί δεν μεταφράζονται σωστά. Ήμουνα πριν από τέσσερι εβδομάδε στην Ουγγαρία και του είπα, κοιτάξτε, αν κάνετε μεταρρύθμιση του συντάγματο ε, που θεωρείτε ότι ε, θα δημιουργήσει προβλήματα, δεν ξέρω, καλύτερα να το μεταφράσετε στα αγγλικά. Γιατί σε εμά η μετάφραση που φτάνει, κανεί δεν μπορεί να την κρίνει κατά πόσο είναι σωστή ή όχι. Και γι' αυτό το λόγο πολλέ φορέ φορές δημιουργούνται παρερμηνίες που είναι περιτές. Δεν λέω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, μπορεί όμως να συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να επισημάνω ότι εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάσω κάτι που να αφορά την Ουγγαρία. Ίσως λοιπόν μπορείτε ε, να προσλάβετε ή να αναθέσετε σε κάποιον ε, που ξέρει Ουγγρικά και να αναφέρει κάτι από τις Ουγγρικές εφημερίδες. Δεν είναι απαραίτητα να είναι κυβερνητικές εφημερίδες. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα εφημερίδων που κυκλοφορεί στην Ουγγαρία. Κοιτάξτε όλα αυτά, η πολυμορφία ε, θα με ε, χαροποιούσε πάρα πολύ. Για τα Βαλκάνια σαφώς και έχω και άλλες πηγές. Η Ουγγαρία πάντως μου είναι πιο σημαντική. Έχετε καμία απορία. Αν όχι θα δώσω το λόγο στον κύριο. Με τα μαύρα μαλλιά, και τα μακριά που τον διέκοψα. Κοιτάξτε, Όσον αφορά τις ε, σκανδιναβικές χώρες, οι χώρες που δεν καλύπτονται, έχουμε ένα πρόγραμμα ε, το οποίο όπως είπαμε ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια και σιγά σιγά επεκτείνεται όλο και περισσότερο ε, με τη βοήθεια που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος μας βέβαια είναι να επεκταθούμε το των δυνατών, κυρίω σε χώρες οι οποίες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία λόγω των εξελίξεων. Και βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώς ε, θα μας στηρίξει και η Επιτροπή. Όσον αφορά τώρα τις εικόνες, ε, τα βίντεο, ε, καλύτερα να σας ενημερώσει ο Ερίκ γι' αυτό. Αλλά σίγουρα η εικόνα είναι πολύ σημαντική για την επικοινωνία μας, κυρίως την επικοινωνία με τους νέους και εκεί έχουμε την πρόθεση να, πρόθεση να επεκταθούμε αλλά όπως σας είπα η εικόνα πολύ απλά κοστίζει περισσότερο και ε, θα πρέπει τουλάχιστον προς το παρόν να περιστούμε στα άρθρα που μεταφράζονται. Για τις εκλογές του 2014 πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ένα εργαλείο όπως η Press Europe μπορεί πράγματι να είναι κάτι το οποίο κατ' ουσίαν ε, στηρίζει την έκθεση των εκπροσώπων σε πάρα πολλές πρωτεύουσες Ευρώπης. Το Press Europa είναι ένα εγχείρημα των ε, συντακτών ε, πολύ σημαντικό πάντα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με το ότι μπορούν να προβληθούν διαφορετικές απόψεις έτσι ώστε η απάθεια, η επιφυλακτικότητα που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, αυτά να καταπολεμηθούν με την ενημέρωση, με τη συζήτηση, να μην είναι κάτι που να παραμένει στην τύχη του. Κατόπιν τούτου θεωρούμε ότι το να χρησιμοποιείται ένα ε, πανευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο είναι σε θέση να προβάλλει διαφορετικές απόψεις, ακόμα και σε χώρους οι οποίοι δεν παίζουν σημαντικό ρόλο αλλά ε, χώρες οι οποίες είναι καθοριστική σημασία, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Ελλάδα, να προβάλλονται διαφορετικές απόψεις ή να γνωρίζει κανείς ε, τι πιστεύουν ε, οι χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία σε σχέση με την Κύπρο και την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Για τα άλλα θέματα που έχουν σχέση με την σύνταξη θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ερικ Μωρίς, ο οποίος μπορεί και να σας απαντήσει. Με συγχωρείτε, όχι εσείς τον δίνετε, εγώ το δίνω το λόγο. Εγώ είμαι η πρόεδρος. Κύριε Μωρίς, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για να απαντήσω στην ερώτησή σας για τον τρόπο με τον οποίο εμείς μπορούμε να ε, προωθήσουμε αυτά τα οποία ε, γράφονται στην Ουγγαρία. Ουσιαστικά, εμείς καλύπτουμε τις 27 χώρες της Ένωσης, αλλά και χώρες υποένταξη όπως είναι η Κροατία, η Τουρκία ή η Μακεδονία. Με την ΕΠ Σάμπατσακ, την ΕΠ Σαμπακ της Ουγγαρίας, ε, τις εφημερίδες αυτές, ε, είχαμε μια συνεργασία. Έχουμε δημοσιεύσει ε, άρθρα τους και δημοσιεύσαμε και άρθρα μιας φιλοκυβερνητικής εφημερίδας. Ουσιαστικά το 63, το 73% των ε, αναγνωστών μας μας διαβάζουν στη μητρική τους γλώσσα. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε μία ε, παρουσίαση του τύπου γενικώ. Για τη Σκανδιναβία, ε, ναι, ότι την ξεχνάμε, σίγουρα είναι κρίμα για τις κλασικές ικανότητες των Σκανδιναβών πρέπει να, κάνουμε, να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των μεγάλων και πλέον ομιλούμενων ιστορικών γλωσσών της Ένωσης και να εξορροπήσουμε με γλώσσες όπως Ρουμάνικα, Τσέχικα, Πολωνικά πρόσφατα έγιναν μέλη της Ένωσης, σχετικά πρόσφατα και τα κριτήρια επιλογής μας είναι ότι οι Σκανδιναβοί μιλάνε πολύ καλύτερα αγγλικά ή γερμανικά για παράδειγμα, άρα έχουν πρόσβαση πολύ πιο εύκολα ε, στον ξενόγλωσσο τύπο και στο ίντερνετ. Το να έχουμε λοιπόν μια τσεχική πολωνική εκδοχή μπήκε ως προτεραιότητα για να μπορούμε να καλύψουμε στον τον περισσότερους Ευρωπαίους σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν. Τώρα, για την εικόνα, για το Press Europe. Εδώ και τέσσερα χρόνια πράγματι έχουμε βελτιώσει τη δυνατότητά μας ε, να αναζητούμε άρθρα σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και για γλώσσες που δεν εκπροσωπούνται στο site μας, άρα αυτό απαιτεί κάποια προσπάθεια. Τώρα έχουμε αντιληφθεί τις μεταλλάξεις αλλαγές των διαδικτυακών εργαλείων και θα προσπαθήσουμε online τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε το λεγόμενο web ντοκιμαντέρ διαδικτυακά ντοκιμαντέρ Θέλουμε να συνάψουμε και εταιρικέ σχέσεις για να μεταδίδουμε ρεπορτάζ. Βέβαια υπάρχει πάντοτε ο περισμός και ανησυχία, η μνά μας αν θέλετε, να δίνουμε πρόσβαση σε αυτά τα βίντεο, σε αυτές τις εικόνες, σε 10 γλώσσες, με την ποιότητα της μετάβασης που έχουμε στο γραπτό περιεχόμενο. Πολύ ωραία. Υπάρχει καμιά ερώτηση ακόμη, όχι. Α, παρακαλώ κύριε Μπόρις. Έρχεσαι τελευταίος και θέλετε να κάνετε και ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ η παρουσίασή σας. Ουσιαστικά σχετίζεται και με το προηγούμενο θέμα μας που ήταν ε, οι γλώσσες ως εργαλείο επικοινωνίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των γλωσσών. Είναι σημαντικό και το έργο σας. Χρήσιμο γιατί αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να συλλέξετε σε μια πλατφόρμα όλες τις σημαντικές ειδήσει και πληροφορίες. Και βέβαια με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο, παρουσιάζοντας δηλαδή τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Βέβαια πρέπει να βρεθεί και χρυσή τομή, γιατί μπορεί ε, σε κάθε χώρα να υπάρχουν ε, κάποια ε, μέσα ενημέρωση που πρόσκειται στην αριστερά, στην δεξιά πρέπει να βρείτε μια ισορροπία. Διαβάζοντας την πολωνική εκδοχή. Ε, πρέπει να σας πω ότι είμαστε η Πολωνία ένα καλό παράδειγμα ενός φαινομένου. Ε, αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη και στον κόσμο δύσκολα ε, μπορούν τα πολωνικά μέσα να τα περιγράψουν, να τα μεταδώσουν, ιδίω ό,τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιορίζονται στο τι συμβαίνει στις ε, συνόδους Κορυφή, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια για παράδειγμα. Πρέπει όμως να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος, να ενημερωθούν σωστά οι συμπολίτες μας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι συνήθω εστιάζουν τα μέσα στην εσωτερική επικαιρότητα και αυτό βέβαια φυσιολογικό είναι. Εσείς κάνετε καταπληκτική δουλειά, νομίζω όμως ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να ευαισθητοποιηθούν οι Πολωνοί, οι Έλληνε, οι Ιταλοί, να καταλάβουν ότι υπάρχεται ουσιαστικά να κάνετε πιο προβεβλημένη και πιο δημοφιλή τη δουλειά σας στα κράτη-μέλη, ώστε η πλατφόρμα σας να είναι ένα είδος ε, υποχρεωτικού περάσματος. Ε, δηλαδή να μπαίνουν σχεδόν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα σας οι πολίτες για να ενημερώνονται. Το θέμα λοιπόν είναι η επικοινωνία πώς θέλετε στα, ε, και στον τοπικό τύπο να ε, έχετε κάποια απορρόφηση και εκεί, γιατί είναι και αυτό δύσκολο. Κοιτάξτε, θα απαντήσω εγώ. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ όλους για τα συγχαρητήρια που έδωσαν στην Press Europe. Είναι σίγουρο ότι πρόκειται για μοναδική εμπειρία. Βλέπουμε τα τελικά αποτελέσματα, αλλά από πλευράς επιμελητίας κρύβονται πίσω από αυτά τα αποτελέσματα ε, πολλοί άνθρωποι και σκληρή δουλειά. Χάρη στην ε, συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μπορέσαμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα χάρη στους Ευρωπαίους φορολογουμένους έχουμε πλέον ε, προβάλλουμε απόψεις για τις οποίες ε, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Έχουμε εξασφαλίσει πρόσβαση ε, στις περισσότερες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσβαση σε πολυάριθμες πηγές πληροφόρησης. Ε, όλα αυτά συνέβησαν προφανώς σταδιακά και καθημερινά προσθέτουμε νέα στοιχεία, τα οποία όμως επισύρουν και νέες δαπάνες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, λέγοντας ότι 90% της κατανάλωσης περιεχομένου ε, συνίσταται σε εικόνες. Το 90% ε, της πληροφόρησης το λαμβάνουμε μέσα από οθόνες, από εφηή τηλέφωνα, από ταμπλέτες, από ε, επιτραπέζιους υπολογιστές, φορτούς υπολογιστές, ε, μπορούμε να προσφέρουμε μια νέα προστιθέμενη αξία γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση των νέων. Γνωρίζετε πώς λειτουργεί το σύστημα και θα τονίσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη διάσταση της δραστηριότητάς μας. Επιθυμούμε επίσης να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση σε τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή. Νομίζω ότι η Κομισιόν δεν έχει στείλει εκπρόσωπο ή κάνω λάθο. Μήπω υπάρχει κάποιο που θέλει παρόλα αυτά να λάβει το λόγο. Από ό,τι βλέπω όμω όχι. Α μην λάβετε το λόγο, τα λεφτά να δώσετε και φτάνει. Μιλήσατε λοιπόν όλοι, παρότι κατ' ουσία μόνο δύο είχαν δικαίωμα να μιλήσουν. Ε, εν πάση περιπτώσει, εγώ χαίρομαι που ήρθατε. Ε, αυτοί λοιπόν που βρίσκονται εδώ θέλω να ελπίζω ότι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές. Ελπίζω αύριο να ανοίξω το δικό σας το έντυπο και να διαβάσω πράγματα ε, που δεν ήξερα γιατί αυτό ε, διευρύνει τον ορίζοντα ανεξάρτητα με την ηλικία του καθενός. Τώρα κλείνει η συνεδρίαση και ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Όσοι δεν είναι συντονιστές, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, να φύγετε.